Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινούμε. Το προσεχές θέμα στην ημερήσια μας διάταξη. Ανακοινώσει του Προέδρου, οι οποίες σχετίζονται προφανώς με τις αποφάσεις των συντονιστών και τη συνεδριάσεως του Ιουλίου και της χθεσινής. Από τους συντονιστές λοιπόν και τη συνεδρίασή τους του Ιουλίου. Η κατανομή των εκθέσεων, ε, αναφορά πλοίων ε, ελιμενιζομένων και αποχωρούντων από... στο ΕΛΚ. Στους σοσιαλιστές η επόμενη έκθεση, με συγχωρείτε Ευρωπαίοι Δημοκράτες ε, σοσιαλιστές, δυσκολεύομαι να συνηθίσω το καινούριο όνομα της ομάδας. Η πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη μια συμφωνία αερομεταφορών με τι ΗΠΑ και την Ισλανδία και το βασίλειο της Νορβηγίας. Η απόφαση λοιπόν αυτή είναι σύμφωνη με τα όσα πράξαμε μέχρι τώρα, με την ε, παράδοση που έχουμε μέχρι τώρα και επανα επανεισάγεται, αυτή η συμφωνία. Ήθελα να επισημάνω δε ότι θα πρέπει και οι αντιπρόεδροι να αναλάβουν να παρακολουθήσουν την ανανέωση αυτών των επανερχομένων ε, συμβάσεων, γιατί δεν πρέπει να τα αναλαμβάνει όλα ο Πρόεδρος. Ανακοίνωση της Επιτροπής για τους στρατηγικούς στόχους Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Πολιτική των Μεταφορών στο 2018 ο Πρόεδρος. Αναλαμβάνει την έκθεση. Έκθεση της Επιτροπής για την ανάλυση σοβαρών ε, παραβάσεων στους κανόνες των οδικών μεταφορών και προβλέψει νομοθεσία στα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωση για το μέλλον των μεταφορών Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στις γνωμοδοτήσεις Λευκή Βίβλος Προσαρμογής στις Κλιματολογικές Αλλαγές ΕΛΚ και η ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βαλτική, επίσης το ΕΛΚ. Βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές οι νομοδοτήσεις ε, εξαρτώνται από την έκθεση της κατουσίαν αρμόδιας επιτροπής. Εφόσον λοιπόν η κατουσίαν αρμόδια επιτροπή αναλάβει ή ε, κατανείμει την έκθεση, αυτό δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα γίνει, θα εκπονήσουμε και εμείς γνωμοδότηση. Αυτά από τις συνεδρίες των συντονιστών του Ιουλίου όπως είπα. Η χθεσινή συνεδρίαση των συντονιστών. Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον κύριο Τζόναθαν Σίλερ από τη Γενική Διεύθυνση των Μεταφορών, όπου μιλήσαμε για την, ε, για την ε, συνθήκη για τις μεταφορές με τα Δυτικά Βαλκάνια και έγινε σχετική ενημέρωση όσον αφορά το διορισμό εισηγητών και συντακτών γνωμοδοτήσεων. Κοινοτικέ προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, επαναδιατύπωση πάλι ανατίθεται στον Πρόεδρο, ο οποίος θα το αναθέσει σε κάποιον αντιπρόεδρο. Το ίδιο ισχύει και για τη συμφωνία για συγκεκριμένες πτυχές των αερομεταφορών μεταξύ ε, αεροπορικών υπηρεσιών μάλλον μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Βραζιλίας. Έκθεση σχετική με την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ως προς την υπογραφή συμφωνίας για ορισμένες πτυχές αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ Ευρωπαϊκής κοινότητα και ε, Βραζιλία είναι διαφορετική έκθεση και πάλι ήταν αναλογάνει ο Πρόεδρος και επίσης το e-call, time for deployment, ηλεκτρονική τηλεφωνία ώρα για ανάπτυξη αποφασίστηκε να μην αναλυφθεί δράση προς το παρόν στο θέμα αυτό. Ζητούμε όμως από την κυρία Γένσεν να ενσωματώσει το θέμα αυτό στη δική της έκθεση για το ITS, την κοινωνική πληροφορία. Αυτά λοιπόν. Συνεχίζουν. Με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ε, υλοποίηση των διατάξεων των σχετικών με την οργάνωση του χρόνου εργασίας όσων ασχολούνται στις οδικές μεταφορές όπου θεωρούν οι συντονιστές ότι θα πρέπει να διατυπώσουμε γνωμοδότηση, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από την επιλογή της Επιτροπής των Κοινωνικών Υποθέσεων και Θεμάτων Απασχόλησης. Και πάλι λοιπόν προτείνουμε να διατυπωθεί, να εκπονηθεί γνωμοδότηση, αλλά υπό τον όρο ότι η Κατουσία αρμόδια επιτροπή θα αναλάβει την έκθεση. Για τα άλλα θέματα, αυτό, αυτό ήταν δύο θέματα, ήταν δύο προτάσεις. Ε, για τις άλλες ε, οι συντονιστές προτείνουν να μην αναλάβουμε δράση. Για δε το ε, πάνελ της ΣΤΟΑ. Έχουμε τρεις υποψήφιους αυτή τη στιγμή, για δύο όμως θέσεις. κύριος Χοκ, από το ΕΛΚ, η κυρία Τίτσαο, από τους Σοσιαλιστές, η κυρία Λίχτεμπεργκερ, από τους Πρασίνους. Όπως είπα, μόνο δύο είναι οι θέσεις μας. Άρα θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία τώρα. ώστε να προσδοριστούν οι δύο συνάδελφοι που θα μας εκπροσωπήσουν στο πάνελ της ΤΟΑ. Θέλει κανείς να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό πριν προχωρήσουμε στη λήψη αποφάσεως. Όχι. Δύο είναι οι ψηφοφορίες αν δεν απατώμε, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ του κύριου Κόκ. Ας καταμετρήσουμε. Oh, Ευχαριστώ για την κυρία Τίτσα. Thank you. All those for Mrs. Lichtenberger. Για την κυρία Λίχτεμπεργκερ. Thank you. Any not voting... Υπάρχει κάποιος που απέχει της ψηφοφορίας. Όχι. Δεν χρειάζεται να σας δώσω τα αριθμητικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αλλά είναι σαφές νομίζω ποιο, ποιον είδε τα, την ανάπτυξη των χειρών, ότι οι δύο πρώτοι είναι Κόχ και ε, θα είναι η εκπρόσωπή μας στο πανελτιστικό της ε, ΣΤΟΑ. Ακροάσεις. Έχουμε ζητήσει από τους συντονιστές να κάνουν τις προτάσεις τους ε, για τις ε, ακροάσεις για το 2010 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Θα σας ρωτήσουν λοιπόν οι συντονιστές σας ε, να υποβάλλετε προτάσεις, ιδέες και ασφαλώς θα συνεχιστεί και η παράδοση της προηγούμενης θητείας όπου επισκέψεις αντιπροσωπιών που δεν εξαντλούνται από τις δύο μεγάλες ομάδες θα παραχωρούνται στις μικρότερες. Εάν λοιπόν μία θέση ε, δεν μπορείτε να την ε, ε, χρησιμοποιήσετε, να την εξαντλήσετε, να την απορροφήσετε, θα τη διαθέτετε σε μικρότερη ομάδα. Επίσης έχουμε πρόσκληση από το Ηνωμένο Βασίλειο για επίσκεψη στο τμήμα μελέτης ατυχημάτων στο ΦΑΜΠΡΟ, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για το 2009. Τρεις από το ΕΛΚ, δύο από τους σοσιαλιστές και ένας από τους φιλελεύθερους. Αυτές είναι οι μόνες θέσεις που έχουν μείνει. Για το ΦΑΜΠΡΟ. Ακροάσεις 2009-2010. Για το υπόλοιπο του 2009 δεν προβλέπονται ακροάσεις. Αποφάσισαν όμως οι συντονιστές να ζητήσουν εξωτερική πραγματογνωμοσύνη, ανεξάρτητους πραγματογνώμονες για ε, μια ανεξάρτητη έκθεση ως προς το μέλλον της, ε, των μεταφορών από πανεπιστημιακούς και όχι από εκπροσώπους του κλάδου με καινοτόμες ιδέες και σύντομες παρουσιάσεις, σύντομη ενημέρωση, ένα brainstorming θα λέγαμε, μισή ημέρα εργασίας με πανεπιστημιακούς, ειδικού επιστήμονες που θα μας δώσουν ιδέες για το μέλλον των μεταφορών. Οι δε συντονιστές απεφάσισαν μαζί με τις ακροάσεις να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο στο μέλλον να χρησιμοποιούμε το σύστημα των ε, workshop των εμπειρογνωμόνων, των ειδικών και όχι μόνο την ακρόαση. Και αυτό ως πηγή ενημέρωσης και γνώσεων για τους βουλευτές για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Οι συντονιστέ γνωρίζουν ότι τι προτάσει του για τι ακροάσει για το 2010 πρέπει να τι υποβάλουν έω τι 18 Σεπτεμβρίου. Δεν κοιμηθήκατε ακόμα. Συγγνώμη που μακρολογώ τόσο. Προχωρώ. Επιτροπολογία. Όσοι από εσά ήταν εδώ και στην προηγούμενη θητεία, θα θυμάστε ίσω ότι είχαμε λάβει απόφαση στην Επιτροπή μα δύο από τους συναδέλφους να ασχοληθούν ιδιαίτερα με τα θέματα της επιτροπολογίας και να επανέλθουν για να υποβάλουν τις εκθέσεις τους, την έκθεσή τους στην Επιτροπή μας τα θέματα αυτά. Αποφάσισαν λοιπόν οι συντονιστές να ε, συνεχιστεί το σύστημα αυτό. Δύο επιφορτισμένοι συνάδελφοι και η απόφαση σχετική θα ληφθεί στην προσεχή συνεδρία των συντονιστών. Ποιοι θα είναι αυτοί δηλαδή που θα αναλάβουν την επιτροπολογία. Επιπλέον αυτού η γραμματεία τακτικά θα περιλαμβάνει στο φάκελο που θα σας υποβάλει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ε, ένα newsletter της επιτροπολογίας, ενημέρωση δηλαδή για θέματα επιτροπολογίας που είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα πραστικό ανάγνωσμα για σας και θα σας επιτρέπει στον καθένα σας να ενημερώνετε, να παρακολουθεί τα θέματα της επιτροπολογίας τακτικά. Και αν κάποιο είναι και ειδικό στην επιτροπολογία, παρακαλώ να έρθει να μου την εξηγήσει και εμένα. Αυτό πάντως σκοπεύουμε να κάνουμε για την επιτροπολογία. Επίση, η κυρία Λίχτενμπεργκερ πρότεινε διεξαγωγή συζήτηση στην Επιτροπή ω προ τα θέματα της, των προβλημάτων, καθυστερήσεων ε, και συνεπειών ε, οικονομικών ή χρονικών από τι καθυστερήσει στην επιβίβαση, την ε, ματέωση πτήσεων. Θα μας απασχολήσει, θα απασχολήσει λοιπόν και αυτό στην επόμενη συνεδρία του συντονιστέ. και επίση για την επόμενη συνεδρία μας τον Οκτώβριο έχω καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή τη ΕΜΣΟ, ε, της ε, οργάνωσης για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών να έρθει να μας μιλήσει όπως επίσης και τον εκπρόσωπο της ε, Υπηρεσίας Ασφαλείας των Αερομεταφορών. Άρα θα έχουμε και ε, τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και τους σιδηροδρόμους εντωμεταξύ κλείσει γιατί θα έχουμε συναντήσει τους επικεφαλείς των σχετικών υπηρεσιών, τους διευθυντές. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα της κατάστασης αυτής, να αντιληφθούμε τις διάφορες ε, πτυχές των διαφορών αυτών τύπων μεταφορών και να είμαστε πιο ενημέροι. Συνάδελφοι, αυτά είχα να πω. Έχετε κάτι να προτείνετε, να ζητήσετε, να ρωτήσετε από τις ανακοινώσεις του Προέδρου, κυρία Ιάλα Σαντέρ. <clears throat> Ναι, Πρόεδρε, θέλω να σας υπενθυμίσω απλά ότι στην πρώτη συνάντηση είχα ζητήσει να έρθει στην Επιτροπή μας, δεν θυμάμαι αν ήταν στους συντονιστές ή κάπως, να υπάρξει πάντως μια παρουσία του υπεύθυνου ε, της ε, δομής κατά της πειρατείας ε, των υπευθύνων τέλος πάντων των Ευρωπαίων υπευθύνων κατά της πειρασίας στη Σομαλία και αλλού. Θα παρακαλούσα και το επαναλαμβάνω αυτό, να τον καλέσουμε γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα και καλό θα ήταν να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, το συμφωνήσαμε και τους προσεγγίσαμε για να μιλήσουμε μαζί τους. Αλλά ξέρετε, οι στρατιωτικοί μερικές φορές ε, δεν είναι εύκολοι να τους βρούμε. Δεν είναι εύκολο να τους βρούμε. Πάντως ε, δεν το ξέχασα. Το έχω βάλει στο ραντάρ του πλοίου μου και έχω ζητήσει από το επιτελείο των, ε, της μονάδας να έρθει να μας μιλήσει. Κάποιος άλλος. Υποθέτω ότι δέχεστε τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Ωραία, ευχαριστώ. Κάναμε και τον ορισμό των εισηγητών. Λοιπόν, προχωρούμε. Ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2010. Συμφωνούμε. Let Να δω και εγώ την κάρτα μου. Έχετε νομίζω τις κάρτες σας, ελπίζω. Αλλιώς πρέπει να πείτε πώς θα ψηφίσετε. Εντάξει. Vote on the section three. Ψηφίζουμε το τρίτο τμήμα του προπολογισμού. Ο κύριος Κόχλιτσεκ είναι ο εισηγητής. Τροπολογία 6438. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ. Καλά, ας κάνουμε ένα τεστ πρώτα. Όσοι θέλετε να κάνετε μια δοκιμή, βάλτε το δάχτυλό σε το δίκτυ, δείτε αν δουλεύει ο δείκτης κλπ. Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. πάρα πολύ ΕΛΚ, περισσότερο από όσοι πρέπει. Ε, τα, οι, πα, οι παλιέ δύσκολα φεύγουν. Και λέγαμε όλα θα αλλάξουν τώρα που έφυγε ο Γκέοργ. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορία. Right, everybody happy. Εντάξει, είστε ικανοποιημένοι όλοι. Ξεκινούμε ουσιαστικά. Μείον 2 ΕΛΚ. Πρώτη τροπολογία. 64-38 της κυρίας Τιτσάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, δεκτή. 64-00 Κράμερ και Ζήλε. Ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα. Για τα ποσά. Πρώτα. Πρόεδρε, ξέρω ότι καθυστέρησα λίγο να έρθω, αλλά έχω την εξή ερώτηση. Δέχονται οι συνάδελφοι να κάνουμε μία δεύτερη χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα, δηλαδή για τις παρατηρήσεις, για να μπορέσουμε να διαγράψουμε ένα κομμάτι, να λέμε δηλαδή σε σχέση με τα δίκτυα, να αφήσουμε έξω τα παραδείγματα, να τα διαγράψουμε και να προχωρήσουμε στα ποδήλατα και τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές, τα σιδηροδρομικά ταξίδια. Και να το δούμε αυτό μετά στα παραδείγματα, διότι, στις παρατηρήσεις, συγγνώμη, διότι θεωρώ ότι το να δίνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ε, μας ε, γεννά πολλές δυσκολίες. Μας περιορίζει δηλαδή περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε. Ίσως λοιπόν αργότερα μέσα παρατηρήσει να μπορούμε να το εισαγάγουμε. Ο Πρόεδρος. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγώ το δέχομαι. Εντάξει. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, Μίκαελ, κύριε Κράμερ. Ναι, το πρόβλημα όμως είναι ότι πάντοτε επισημαίνεται ότι πάνε μαζί τα δύο αυτά συστήματα, το Eurovelo και η σιδηρόδρομη Και νομίζω ότι δεν ε, μπορούμε να τα διαγράψουμε και τα δύο. Το έχουμε αποφασίσει όλοι τους ή άλλους. Επειδή πάντοτε λέγεται ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, αυτό θέλουμε να μπει μέσα στο κείμενο. Ναι, αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα. Πρόκειται για τον τουρισμό σε τελευταία ανάλυση και εδώ επανέρχομαι και στην παρατήρηση που κάναμε και χθε σχέση με τη διάκριση μεταξύ μεταφορών και τουρισμού. Τουρισμός είναι εδώ. Εμένα δεν ε, με ενοχλεί να παραμείνει η, αίρια, η έννοια Eurovelo ως και αυτή μέσα στο κείμενο, αλλά χωρίς συγκεκριμένα παραδείγματα. Το δέχεστε? Έτσι θα κάνουμε. 64.00 λοιπόν. Πρώτο τμήμα. Προπαρασκευαστικέ δράσει βιώσιμου τουρισμού υπέρ. Κατά. αποχέ. Δεκτό τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Είχα ζητήσει, υπήρχε χωριστή ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα των παρατηρήσεων και νομίζω θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα το σιδηρό παραπέτασμα και μετά τις παρατηρήσεις χωρίς τον όρο σιδηρού παραπέτασμα. Κύριε Γιάλα στην τροπολογία όπως ε, εμφανίζεται. Αυτό που έκανε ο κύριος Κράμερ είναι να βγάλει το γιουροβέλο και να βάλει απλά και μόνο το παράδειγμα του σιδηρού παραπετάσματος. Εγώ τι λέω. Λέω ότι καταψηφίζοντας την τροπολογία στις παρατηρήσεις του κυρίου Κράμερ παραμένει να παραμείνει το γιουροβελό, δηλαδή ε, δίκτυα ποδηλατικών διαδρομών όπως το, ε, το γιουροβελό. Στα ισπανικά τουλάχιστον η τροπολογία αυτό που ε, βλέπω είναι ότι ο κ. Κράμερ έβγαλε το παράδειγμα του Eurovelo και έβαλε αποκλειστικά το ε, δρόμο που, στα ίχνη του σιδηρού παραπετάσματος, τη διαδρομή στα ίχνη του, του σιδηρού παραπετάσματος. Εγώ πιστεύω ότι αν καταψηφίσουμε τις, τροπο, τις ε, τροπολογίες Κράμερ στις παρατηρήσεις, ανακτούμε και τα δίκτυα αποδηλωτικών διαδρομών και το Eurovelo. Αυτό νομίζω. Καλά ξεκινάμε. Καλά ξεκινάμε. Πρώτη ψηφοφορία. Ε, δώστε μου λίγο χρόνο να το τσεκάρω. Right, Michael, do you agree to... Μίχαελ, συμφωνείς με το αίτημα του κύριου Γκρός αν ναι, θα υπάρξει χωριστή ψηφοφορία. Αλλιώ, όχι. Μίχαελ. Η κυρία, Φρα... Ε, κυρία Ιάλα με έχει καταλάβει λάθος νομίζω. Η γραμμή αυτή του σιδηρού παραπετάσματος, τα ίχνη του σιδηρού παραπετάσματος είναι κομμάτι του γύρω βέλο. Γιατί λοιπόν να στρέφεται κατά αυτής της έννοιας σε τελευταία ανάλυση ε, εορτάζουμε και την 20η επέτειο της κατάρρευσης του συντήρου παντραπετάσματος. Άρα δέχεστε την πρόταση για χωριστή ψηφορία, κύριε Κράμερ, σωστά, σωστά. So Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα των παρατηρήσεων. Μπορείτε να μας το διαβάσετε. Γιατί είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ψηφίζουμε. Θέλετε να με ακούτε ή όχι, λέει. Θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας ως πρόεδρος. Τέλος πάντων, θα το προσπαθήσω. Κύριε Γκρός. Πρόεδρε, για να διευκολύνω τη συνάδελφα. Ή τους συναδέλφους καλύτερα. Μήπως το σιδηρούν παραπέτασμα, τα ίχνη του σιδηρού παραπετάσματος, να ήταν καλύτερο να τα ψηφίσουμε χωριστά. Και αν δεν μείνουν μέσα στο κείμενο, μπορούμε να ψηφίσουμε τις παρατηρήσεις χωρίς τις τρεις αυτές λέξεις ε, σε ένα χωριστό κείμενο. Πέντε λέξεις. Νομίζω ότι το έχει περιπλέκει πολύ κατάσταση περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Περιμένω ένα λεπτό να το τσεκάρει και ο συντάκτης της τροπολογίας. Λοιπόν, ψηφίζουμε καταρχήν τις λέξεις στα ίχνη του σιδηρού παραπετάσματος. Ποιοι είναι υπέρ της συμπερίληψης στο κείμενο αυτών των λέξεων. Κατά. Αποχές. Πάβουν να υπάρχουν. Το λοιπό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Και έλεγα να πω να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ τώρα, κάνα κάνα αλλά τέλος πάντων. Τροπολογία 6439, τι κάου, υπέρ κατά αποχές δεκτή 64.00 του 64.01 συγγνώμη του εισηγητή και 64.40 και 64.40 της κυρίας Αγιάδας που είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές ας κάνουμε έναν έλεγχο ηλεκτρονικό Ψηφίσατε. Πέρα ψηφοφορία. 23 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή. Δεκτή. Επόμενη τροπολογία. 6402 του εισηγητή για την ε, δορυφορική πλοήγηση της, ΟΥΠΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6405 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές δεκτή 6407 του εισηγητού υπέρ παρακαλώ κατά αποχές υιοθετείται προφορική υδροπολογία επιχειρή όχι. Όχι. Συγητή, κύριε Κόντσεκ. Πρόεδρε, ο κύριο Φιλίππη ανέφερε πω, ε, εάν όταν έρθουν εδώ στα εταιρείε και εφόσον αυτή τη στιγμή του δίνουμε χρήματα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πω να εξασφαλίσουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δημιουργίες νέων θέσεων. Και αν δείτε πραγματικά στο παράρτημα της, του ελέγχου ψηφοφορίας, του καταλόγου ψηφοφορίας θα δείτε πως υπάρχουν οι ατομικές θέσεις οι οποίες αναφέρονται στην κατανομή που γίνεται όσον αφορά τις εταιρείε αυτά. Εάν θέλουμε λοιπόν, εφόσον τους δίνουμε πρόσθετα χρήματα και στην ΕΑΣΑ όλα αυτά τα χρήματα συνδέονται με ειδικέ απασχολήσεις και πρέπει να διασφαλίσουμε πως αυτά τα, αυτές οι θέσεις εργασίες, αυτές οι απασχολήσεις αυξάνονται. Ε, ο, ο κ. μίλησε χθε κατά αυτής της απόψεως και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε πως πολλές απασχολήσεις είναι περιορισμένες στις εργασίες, περιορισμένες. Και παράδειγμα, νέα ΣΑΠ έτσι υπήρξαν, αλλά όχι πάρα πολλέ. Υπήρξαν λοιπόν περισσότερα χρήματα, αλλά όχι περισσότερε θέσει εργασία. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο έρχεται αυτή η προφορική προφολογία και κατατίθεται μέσα σε αυτόν κατάλογο των τροπολογιών. Στο παράρτημα επίση θα δούμε ποιε είναι οι δικέ μα θέσει. Εάν θέλετε, μπορείτε και επιμένετε, μπορώ να σα διαβάσω αυτό ναι. Ναι, Πρόεδρε. Νομίζω ο κ. Μπράμπερ μίλησε χθε κατά, κατά της αύξησης και των θέσεων εργασίας σε αυτές τις εταιρείε, αλλά η εξήγηση της Κομισιόν υπήρξε ότι εάν θέλετε να βάλετε περισσότερα χρήματα θα πρέπει να έχετε και νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ο σκοπός της τροπολογίας η οποία παρουσιάζεται σήμερα σαν προφορική ενώπιόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, θα το εξετάσουμε κατηδίαν και κάθε φορά πραγματικά που έρχεται ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τα διάφορα για τις Προφορική λοιπόν τροπολογία ε, που γυρίθηκε από, τον εισηγητή. Ως παρακαλώ της προφορικής τροπολογίας κατά υιοθετείτε. υιοθετείται 64-10 ο εισηγητής είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. όχι προφορική τροπολογία πάλι Πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε την προφορική. Την προφορική ξανά. Από τον κύριο Κόλιτσεκ, Τσέκος είναι υπέρ παρακαλώ της προφορικής, κατά Αποχές υιοθετείται. 64-46, Τσάου ο συγητής, παρακαλώ. Εάν το προηγούμενο ε, έχει υιοθετηθεί το δικό μας αυτό το 6446 καταπίπτει διότι είναι προσθήκη αυτή. Θα πρέπει να το θέσουμε βεβαίω σε, σε ψηφοφορία. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να ληφθεί ως προσθήκη. 64-46 τικάου, τικάου, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64-12 του εισηγητού συνυπέρ παρακαλώ κατά αποχές υιοθετείται ε, 64-44 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 64-16 όσοι είναι υπέρ παρακαλώ θα μπει αυτό μόνο στις παρατήσεις κατά αποχές υιοθετείται 64-17 Γέντσεν Γκρίσμπεκ όσοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. Ένας ή δύο περισσότερο είναι στο ΕΛΚ. Ωραία. Εντάξει, το ελέγξατε. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν 38, 20 υπέρ, 17 κατά, μία αποχή υιοθετειτε 6415 του εισηγητού καταπίπτει. Καθώς και άλλα. Πάμε στο 6419 19 Κατέπεσαν όλα τα προηγούμενα. Του εισηγητού πάλι περ κατά, αποχές. Υιοθετείτε. 4.20 του εισηγητού, ο συνυπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Όλες οι υπόλοιπε, α, ε, συγγνώμη, η, προσ, η προφορική προτροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε 6424 του κυρίου Κράμερ, ε, ψηφοφορία σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχουν μόνο τα ποσά, ως είναι υπέρ των ποσών, κατά, αποχές, υιοθετείται. Δεύτερο μέρος είναι οι παρατηρήσεις. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Και τρίτο μέρος είναι η διαγραφή της περιβόητης λέξης ε, σιδηρού παραπέτασμα υπέρ, κατά, αποχές Υιοθετείτε. Το 6422 του εισηγητού καταπίπτει. Ο επίσης του Γένσεν και των υπολείπων. Και πάμε στο 6425 του εισηγητού πάλι. Ο εισηγητής υπέρ είναι κατά. Αποχές υιοθετείται. 6426 του κυρίου Κράμερ, τιματική ψηφοφορία. Όσοι είναι υπέρ των ποσών, δύο μέρη, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Δεύτερο μέρος οι παρατηρήσεις, όσοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Το 6453 καταπίπτει. 6454, Αλβάρε, Αγιάλα Σέντερ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, υιοθετειτε 6455 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 6429 του κ. Κόκ, τιματική ψηφοφορία, ποσά και παρατηρήσει στα δύο μέρη. Το πρώτο μέρο, ποσά, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, υιοθετείτε. Παρατηρήσει το δεύτερο μέρο, υπέρ. Κατά. Αποχές, η ίδια πλειοψηφία και υιοθετείται κατά τον αυτό τρόπο. 64-56, 56 γνωμη καταπίπτει. 64-32 της κυρίας Γιάννης ενώ είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. 64-32 της κυρίας Γιάννης έλεγχος ηλεκτρονικός. της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 39, 21 υπέρ, 18 κατά, καμία αποχή. Υιοθετείται. 64-33 της κυρίας Γέντσεν, όσοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 64-57 της κυρία Τιτσάου, τμηματική ψηφοφορία ε, ποσά και παρατηρήσεις στα δύο τμήματα. Το πρώτο μέρος είναι τα ποσά, ως είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απερίφθη Το δεύτερο μέρος οι παρατηρήσεις, ως είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απεριφθεί. 64-58 της κυρία Τσάου είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές 6434 του εισηγητού, ως είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απερίφθη. όχι υιοθετείτε λέει ο πρόεδρος υιοθετείτε προφορική τροπολογία ως είναι υπέρ κατά αποχές 6460. Κύριε Αλβάρες και Αγία σεντερος Σέντερος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 64-61. Κυρία Αλβάρες οι ίδιοι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 64-62. Οι αυτοί πάλι συντάξαντες υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 6436, ο κύριος Κράμερ, ο κύριος Ζήλε θεματική ψηφοφορία έχετε τρία μέρη τα ποσά οι παρατηρήσεις και διαγραφή της, λέ, της λέξεως ε, στηρούν παραπέτασμα πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε παρατηρήσεις δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα ψηφίστε παρακαλώ δεύτερο μέρος είναι οι παρατηρήσεις τις οποίες ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή ψήφισαν οι πάντες πέρας ψηφοφορίας ψηφίσαντε 40 18 υπέρ 21 κατά μία αποχή απερίφθη το δεύτερο μέρος και πάμε στο τρίτο μέρος Ναι, δεν υπάρχει λόγο να το ψηφίσουμε γιατί το απορρίψαμε και την προηγούμενη φορά. Ο κύριε παρακαλώ. Πρόεδρε, γι' αυτό το λόγο θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι στην τροπολογία, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, που έχει την ίδια διατύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, όπου δεν είχαμε κάνει δεκτές τις παρατηρήσεις και πάλι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για το συντηρούν παραπέτασμα. Δηλαδή να παραμείνει το αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής ψηφοφορίας για τις παρατηρήσεις και να μην γίνει ψηφοφορία για το συντηρούν παραπέτασμα. Έτσι δεν είναι. Έχετε δίκιο πραγματικά. Ο κύριος Κόλιτσεκ έχει το λόγο εισηγητής παρακαλώ. Νομίζω πως πρέπει να ενοποιήσουμε τις τέσσερις αυτές περιπτώσεις και όλες τις, τα ποσά και τις παρατηρήσεις οι οποίες θα, θα συσσωματωθούν αυτές, θα συγκεντρωθούν. Άρα, ερχόμαστε στο 64-36 του κυρίου Κράμερ και Ζήλε. Υπάρχει σημαντική ψηφοφορία, ρωτάει. Ναι, Δύο μέρη, ποσά, παρατηρήσεις, ερωτηματική, τα ποσά πρώτον υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Παρατηρήσει υπέρ, δεύτερο μέρος, κατά, αποχές, απερίφθησαν. 64-37 της κυρίας Γέντσεν, υπέρ παρακαλώ, κατά, να ελεγχθεί καλύτερα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, πάρτε τις κάρτες σας. 64-37. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. ψηφισαν 40, 24 υπέρ, 16 κατά. 40 ψήφισαν και αυτό είναι σωστός αριθμός. Τώρα. Ε, στις προτάσεις. Ένα Αλβάρες Αγιάλα Σέντερ ο είναι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. δύο. Κύριο Κράμερ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. τρία. Αλβάρες. Αγερασέντερο. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. τέσσερα. Για αυτή η συντάξη υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Πέντε, κυρία Γέντσεν υπέρ παρακαλώ κατά αποχές υιοθετείτε. τελική ολική ψηφοφορία στο σύνολό της δηλαδή άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ ψήφισαν οι πάντες Πέρας. Ψήφισαν 40, 40 υπέρ, 0, 0. Πλήρης ομοφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή τη και γραμματεία επίση, η οποία βοήθησε πάρα πολύ τον πρόεδρο σε αυτή τη δύσκολη αποστολή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επόμενο σημείο η Σουηδική Προεδρία λίγα λεπτά αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επανέλθουμε τη Σουηδική Προεδρία. Ευχαριστώ.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 Συνάδελφοι, θα ήθελα να, καλωσορίσω την Υπουργό Μεταφορών και Τουρισμού της Σουηδίας για τις επικοινωνίες κυρία Τόρσεν δεν μπορώ να πω καλά το όνομά τους είναι βεβαίω αυτή η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και έχουμε αυτή τη στιγμή το προνόμιο να την υποδεχθούμε χθε και να έχουμε μαζί της ένα δείπνο χθε το βράδυ και βεβαίως είστε η πρώτη από την Προεδρία η οποία έρχεστε ενώπιον της Επιτροπής Τουρισμού Μεταφορών και Τουρισμού και πιστεύω πως πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι εκτιμούν ιδιαίτερα τη δική σας παρουσία εδώ. Ευχαριστώ λοιπόν Υπουργέ που είστε εδώ και σας δίνω με σωστό λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να σας συγχαρώ όλους σας για την εκλογή σας ως μέλη του Κοινοβουλίου και ως, ε, για την τοποθέτηση στην Επιτροπή αυτή. Και εγώ και η Προεδρία μας θέλουμε να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και μεγάλη επιτυχία στη νέα θητεία σας. Η πρόθεσή μας είναι μαζί με σας να κλείσουμε τα θέματα μεταφορών που βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή και θα παρουσιάσω σύντομα τις κύριες προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών. Και αν χρειαστεί θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα όταν απαντώ στις ε, ερωτήσεις σας. Ξέρω ότι τώρα μόλις ξεκινάτε ε, τις δουλειές σας και πολλοί εισηγητές δεν έχουν ακόμα ε, οριστεί. Είμαι ωστόσο πεπισμένος ότι θα έχουμε πολλές δυνατότητες να συζητήσουμε με καρποφόρο τρόπο κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας αντιμετωπίζει δύο προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε εξαιρετικά σοβαρά. Πρώτα πρώτα την οικονομική κρίση και κατόπιν την αλλαγή του κλίματος. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να δούμε την ε, πολιτική μεταφορών εκτενέστερος ε, λύση για σημαντικά ζητήματα ε, για την δημιουργία μιας οικολογικά αποδοτικής οικονομίας. Το, σύστημα μεταφορών είναι αγκαίο για τη διατήρηση της ευημερία στην Ευρώπη και για την ανταγωνιστικότητά μας. Και ο σχεδιασμός της πολιτικής μεταφορών είναι ένα βασικό στοιχείο αν θέλουμε να πετύχουμε ε, ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. Ήδη πέρυσι η Σουηδία μαζί με την Τσεχία και τη Γαλλία έθεσαν τις προτεραιότητες μέσα σε ένα 18 μήνο πρόγραμμα πλαίσιο και είχαμε συμφωνήσει να αντιμετωπίσουμε τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, βιώσιμες και ανταγωνιστικές μεταφορές. Δεύτερον, ασφαλά, ασφαλή μέσα μεταφορών και τρίτον την ανάπτυξη ενό έξυπνου συστήματο μεταφορών. αυτέ τι προτεραιότητε τι συνεχίζουμε σαν Σουηδική Προεδρία. Ε, σίγουρα τα επόμενα χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το πρόβλημα του κλίματο. Εμεί θέλουμε να επιτευχθεί συμφωνία στην Κοπενχάγη το Δεκέμβριο αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητά τη ε, σύμφωνα με την ε, στρατηγική της Λισαβόνας και να μην ξεχάσουμε τα σημαντικά ζητήματα της, ε, του περιβάλλοντος ε, και της ασφάλειας των μεταφορών. Κατά άποψή μου, μια, ένα, ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών μακροπρόθεσμα έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης και μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση οικονομίας το σύστημα μεταφορών είναι, του, είναι τμήμα του προβλήματος ε, του κλίματος αλλά και τμήμα της λύσης τους. Κατά την άποψή μου, μείωση, η μείωση των ε, ε, εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί με μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές και με πιο αποτελεσματικές μεταφορές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ενιαίο σύστημα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι 27 συστήματα. Για να μην πω 108 ε, δεδομένου του ότι πολλές χώρες έχουν διαφορετικά συστήματα για τα διάφορα διαφορετικές ε, τεχνικές για τα διάφορα είδη μεταφορών. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ε, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργία των συστημάτων μεταφορών. Για το λόγο αυτό η Σουηδική Προεδρία θα θέσει τρεις προτεραιότητες. Την πολιτική μεταφορών της Ένωσης μετά το 2010, την αποτελεσματική επιμελητία για τις μεταφορές ε, και το έξυπνο σύστημα μεταφορών, το ITS. Θα δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα στο μέλλον των μεταφορών. Το 2001 η Επιτροπή υπέβαλε μια λευκή βιούλο για την ε, ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών μέχρι το 2010 και τώρα που τελειώνει αυτή η δεκαετή περίοδο θα πρέπει να επεξετάσουμε το σύστημα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη νέα ανακοίνωση τη Επιτροπή με τίτλο Ένα βιώσιμο μέλλον των μεταφορών. Θα ήθελα εσεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατό μια ε, πυκνή συζήτηση για το μέλλον των ευρωπαϊκών, της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και είναι σημαντικό αυτό να γίνει αυτή τη φορά και με τους χρήστες των συστημάτων μεταφορών, του συστήματος μεταφορών. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη άλλες διαστάσεις, τη γύρανση του πληθυσμού, τη μετανάστευση, την εσωτερική κινητικότητα, τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και βεβαίως την, με, με έμφαση στην, στην έλλειψη ορυκτών καυσίμων και την αστικοποίηση. Η Προεδρία μα θα δώσει μεγάλη σημασία σε αυτή τη σημαντική ανακοίνωση τη Επιτροπή και θα οργανώσουμε μια υπουργική συζήτηση στη συνάντηση του Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών και ενέργεια και θα υιοθετήσουμε σχετικά συμπεράσματα στη συνάντηση του Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να ακούσω και τι δικέ σα απόψει για τι μεταφορέ στο μέλλον και κατά συνέπεια ε, προσβλέπω σε ένα συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ των ε, θεσμών μας. Ένα κοινό σεμινάριο που θα οργανώσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις σχετικά. Οι κοινέ συζητήσει θα, να επιτρέψουν, θα πρέπει να μας επιτρέψουν να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του αντίκτυπου των πολιτικών μεταφορών, ενώ ταυτόχρονα θα θέσουν νέους στόχους και την βέλτιστη μέθοδο για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών που πληρεί τι ε, οικονομικέ, κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ ανάγκε τη κοινωνία απαιτεί να αναπτυχθεί καινοτόμα τεχνολογία και να επιταχυνθεί αυτή η καινοτόμα τεχνολογία. Ελπίδα μας είναι να φτάσουμε σε μια συμφωνία για την πρώτη επιτροπή για το πλαίσιο εισαγωγή ενός έξυπνου συστήματος μεταφορών για τις οδικές μεταφορές που θα μειώνει την ε, συμφόρηση, τις εκπομπές, την ρήπανση και τα χήματα και θα επιτρέψει σε κάθε μορφή μεταφορών να αναπτυχθεί με τον βέλτιστο τρόπο. Οι νέες τεχνολογίες όπως το ITS θα μπορέσουν να παράσχουν ε, αυτούς που χρησιμοποιούν συστήματα μεταφορών με πιο προηγμένες και πιο καλές υπηρεσίες. Τα νέα συστήματα διαχείρισης μεταφορών μπορούν να βοηθήσουν την αύξηση της ε, ε ασφάλειας και να ελπίζω να πετύχουμε συμφωνία σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αναφέρω δύο βασικά, βασικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας. Στις 21 του Σεπτεμβρίου στη Στοκχόλμη ε, θα ξεκινήσει το 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο για έξυπνα συστήματα μεταφορών. Το κύριο θέμα του θα ήταν το ITS στην καθημερινότητα. Επίσης η Προεδρία θα οργανώσει μια συνάντηση ψηλού επίπεδου στο Γκέτεμπουργκ στις 26-27 Οκτωβρίου με τίτλο «Οι οδικές μεταφορές στο μέλλον, ασφαλείς και καθαρές». Ο στόχο τη συνάντηση είναι να δείξει πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν περαιτέρω στην δημιουργία ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον οδικών μεταφορών και θα επιταχύνει την εισαγωγή νέων και γνωστών τεχνολογιών ταυτόχρονα. Κάθε χρόνο περίπου 40.000 άτομα σκοτώνονται ακόμα σε ατυχήματα, σε οδικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα μέχρι να πετύχουμε το στόχο που είχαμε θέσει για 27.000 θύματα ε, το 2010. Η Επιτροπή προετοιμάζει την, το τέταρτο πρόγραμμα, για την ασφα... Ε, πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια για την περίοδο 2010-2020. Για να πετύχουμε τους στόχους πρέπει να δώσουμε έμφαση στους τομείς που παράγουν αποτελέσματα προσαρμογή της, καλύτερη προσαρμογή ε, ταχύτητας, αύξηση της οδήγησης ε, από άτομα που δεν έχουν πιει, ε, χρήση ζωνών ασφάλειας. Στόχος μας είναι στο να πετύχουμε βελτίωση και ταχύτητα, ταχύτητα στην επίτευξη των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, στην ασφάλεια των μεταφορών θα δουλέψουμε αυξάνοντας την ποιότητα των μεταφορών ιδιαίτερα ό,τι αφορά την προσωπική ασφάλεια και την μείωση των ατυχημάτων. Θα εξετάσουμε την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με κοινέ αρχές για την ε, για, την, ε, για τις ε, εισφορές τελών αεροπορικής ασφάλειας σε κοινωτικά αεροδρόμια και την δημιουργία ειδικών, μη διακριτικών, ενός πλαισίου για ειδικά και μη διακριτικά τέτοια αεροπορικά τέλη. Επίσης, θα εξετάσουμε την πρόταση κανονισμού για τα ατυχήματα και τις έρευνες αεροπορικών ατυχημάτων με εναρμονισμένες διαδικασίες σε περιπτώσεις ε, αεροπορικών ατυχημάτων. Ε, τα, ατυχήματα, τα αεροπορικά ατυχήματα των τελευταίων μηνών υπογραμμίζουν τη σημασία μιας τέτοιας πρότασης. Η βελτίωση της ποιότητας των μεταφορών και της προσωπικής ασφάλειας των, αλλά και της προστασίας των δικαιωμάτων των ε, επιβατών είναι βασική, πρέπει να παραμείνουν βασικά τμήματα της πολιτικής μεταφορών της Ένωσης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τα δικαιώματα των ε, επιβατών και να δώσουμε έμφαση στις ανάγκες και τα δικαιώματα των χρηστών των μεταφορών. Δίνουμε λοιπόν μεγάλη σημασία στι δύο προτάσει τη Επιτροπή που έχουν στόχο να ενισχύσουν τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορείο ή με υπεραστικά λεωφορεία, καθώ και διαθαλάσσει ή με εσωτερικέ πλωτέ οδού θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε σε αυτούς παρόμοιες ρυθμίσεις με αυτές για τους χρήστες των σιδηροδρόμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη εξέτασε πρώτη ανάγνωση και τις δύο αυτές προτάσεις και ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, τόσο ώστε όλοι οι επιβάτες να έχουν καλύτερη προστασία όταν υπάρχει καθυστέρηση ή ακύρωση των μεταφορών τους. Και τα κύρια κείμενα αυτά εξασφαλίζουν το ότι άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή με αναπηρία δεν θα αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να πετύχει το στόχο να υλοποιήσει η εσωτερική αγορά στου διάφορους τομείς μεταφορών, τόσο ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τη. Το έργο αυτό, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη απλοποίηση νομοθετικού χαρακτήρα, να μειώσουμε τα περίτα διοικητικά βάρη, ιδίω στον τομέα των σιδεδρόμων και των πλοίων. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που δίνουμε στην ε, οδηγία για την αναφορέ τις αναφορές διατυπώσεων ε, σκαφών που εισέρχονται ή εξέρχονται σε κοινωτικούς λιμένες. Χάρη στην μεγάλη ακτογραμμή της Ευρώπης και το μεγάλο ρυθμό των λιμένων, ο, ο τομέας είναι ένα βασικό εναλλακτικό μέσο στις οδικές μεταφορές. Η εφαρμογή, του... της δημιουργία... και η υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα θα βελτιώσουν την κατάσταση αν απλοποιήσουμε τις διαδικασίες των κλάδων. Ελπίζουμε να υπάρξει γρήγορη συμφωνία με το Κοινοβούλιο στο κείμενο αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο θα ήθελα να αναφερθώ και στην στρατηγική για τη Βαλτική, ένα, μια σημαντική συνολική προτεραιότητα για τη Σουηδία και που αφορά εμπολής και τον τομέα των μεταφορών. Μέσω της οδηγίας για τις διατυπώσεις αναφοράς και την επερχόμενη αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων μπορεί να δημιουργηθούν υποθέσεις για να εφαρμοστεί η στατική αυτή και να έχουμε νέα αποτελεσματικά, νέες αποτελεσματικές λύσεις μεταφορών όπως τις πράσινους διαδρόμους και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα για άλλες περιφέρειες. Στον σιδηροδρομικό τομέα η Ένωση προσπάθησε να δημιουργήσει μια, αγορά, μια αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα λειτουργεί σωστά. Τρία σιδηροδρομικά πακέτα έχουν εγκριθεί από το 2001 για να πετύχουν το στόχο αυτό. Η εμπειρία δείχνει ότι η απελευθέρωση της αγοράς είναι αποτελεσματική και επιτυχής όταν εφαρμόζεται πλήρως. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος και έχουμε μεγάλο δρόμο να κάνουμε πριν πετύχουμε το στόχο μας. Ξεκινώντας, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρω το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο, ούτως ώστε να υπάρχει ένα σιδηροδρομικό σύστημα με εναρμονισμένη δυνατότητα κατανομής ε, χωρητικότητα και πρόσβαση σε τερματικού σταθμού. Ε, η προσπάθειά μα για την απελευθέρωση αυτή συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια τη προεδρίας μα. Ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία μαζί σας για τον κανονισμό για, την, ε, για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών που θα είναι πλήρω προσβάσιμο στην Ευρώπη. Η κοινή θέση για την πρόταση αυτή θα υποβληθεί σε εσά το συντομότερο δυνατό. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών σιδηροδρόμων εμπορευματικών μεταφορών θα επιτρέψει την αύξηση της μεταφοράς, των μεταφορών από τους δρόμους στο σιδηρόδρομο. Η ανάπτυξη ε, δια λειτουργικών τερματικών θα μπορέσει να επιτρέψει ε, την εξέβρεση λύσεων και μια έξυπνη ένταξη όλων των μορφών μεταφοράς στο σύστημα αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μεταφορών επιβατών και φορτίου. Αλλά καλή συνεργασία μεταξύ δομών, των εθνικών δομών και διοικήσεων θα οδηγήσει καλύτερες δυνατές λύσεις πιστεύω. Επίσης, η Σουηδική Προεδρία στόχο έχει την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ως προς την οδηγία για το χρόνο εργασίας για τους οδηγούς φορτηγών στις οδικές μεταφορές. Γνωρίζω ότι αρμόδια κατ' ουσίαν ε, στην υπόθεση αυτή δεν είναι η Επιτροπή των Μεταφορών και Τουρισμού, αλλά η ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Αλλά θα ήθελα να συζητήσω το θέμα μαζί σας ούτως ή άλλως. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις ε, μικρές επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών η πρόταση οδηγίας αυτή. Έχει αλλάξει πολύ ο τομέας των μεταφορών τα τελευταία χρόνια και με πολύ σημαντικές κοινωνικές ε, διαστάσεις. Η προϋποθέσεις λοιπόν για την ε, είσοδο στην αγορά αυτή, στον τομέα αυτών, οδηγεί σε μια όλο και περισσότερο διονγκούμενη γκρίζα ζώνη των λεγόμενων αυτοαπασχολουμένων. Προτείνει λοιπόν από το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την, τον εξυγχρονισμό με την οδηγία 2002 κάθετος 15 του τομέα αυτού με στόχο την απαγόρευση, τον αποκλεισμό του φαινομένου των ε, ψευδός αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Το Συμβούλιο υιοθέτησε γενικές κατευθυντήρε γραμμέ το Μάρτιο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όντως να προχωρήσουμε σύντομα στο τομέα αυτόν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ είναι η οδηγία για την Ευρωβινιέτα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι Υπουργοί των Μεταφορών δύο φορές έχουν εξηγήσει ε, ποιο θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η πρόταση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι από του συναδέλφου μου συμφωνούν με του κυρίου στόχου και τι προτάσει. Υπάρχουν όμως σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες και ε, επιπτώσεις. Και άρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη συζήτηση μέχρι του λάβει το ε, Συμβούλιο μια τελική θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τεχνολογικού τύπου μελέτες για να επιτρέψει τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν καλύτερα τις συνέπειες της πρότασης, πράγμα το οποίο πρώτα θα πρέπει να προηγηθεί της οποιασδήποτε ανάληψης συζητήσεων. Για να συνεχίσω και πάλι στον τομέα του περιβάλλοντο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να υποβάλει πρόταση και μια οδηγία για τι εκπομπέ οξυδίων του αζότου, ε, και πριν από ε, λίγο καιρό πρόταση για την ε, συμπερίληψη, και των εκπομπών από τις αερομεταφορές υιοθετήθηκε έτσι ώστε να μπορέσει να, λάβει η να αναλάβει η Επιτροπή το έργο της και ως προς τις περιβαλλοντικές συνέπειες των αερομεταφορών. Θέλουμε λοιπόν κοινέ διατάξεις για την επιβάρυνση σε εκπομπές αζότου, ε, οξυδίων του αζότου από τα ευρωπαϊκά, σε επίπεδο μάλλον ευρωπαϊκών αεροδρομίων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ε, προωθήσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ε, επικοδομητικά για μια καλύτερη πολιτική των μεταφορών, οικολογικά αποτελεσματική και οικονομική πολιτική των μεταφορών για περισσότερε θέσει εργασία και καλύτερο περιβάλλον. Και πριν κλείσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η νέα νομοθεσία δεν αποτελεί πάντοτε το, την μόνη ή την καλύτερη λύση. Είναι απαραίτητο εξίσου να εξασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία που ήδη ισχύει εφαρμόζεται σωστά. Και εδώ έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Σε ορισμένε περιπτώσει, άλλα μέτρα μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικά και αποτελεσματικά από την ε, ε, εισαγωγή νέας νομοθεσίας. Επί παραδείγματι, στον χώρο της οδικής ασφάλειας, η αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών ε, έχει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την εισαγωγή νέων μέτρων. Η σημασία μιας σωστής τάσης προς τις οδικές μεταφορές ως προ την κίνηση στους δρόμους μας δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Είναι τεράστια. Και εδώ έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κράτη-μέλη τεράστιο ρόλο να διαδραματίσουν. Πρόεδρε, είμαι στη θέση τώρα να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση ενδεχομένω έχετε και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια ολόκληρη τη Σουηδική Προεδρία. Είμαι πάντα σε θέση για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση παρατήρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. και την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ακούσω τώρα πρώτους τους συντονιστές και μετά τους λοιπούς συναδέλφους από την Επιτροπή. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι για να μπορέσει η, προ... κυρία Υπουργό να απαντήσει στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις μας θα πρέπει να τις αφήσουμε αρκετό χρόνο. Θα ξέρετε ότι έχω γίνει δεξιοτέχνης του σφυριού αυτού και όταν βλέπω ότι θα δαπανείτε πολύ χρόνο θα σας σταματώ. Παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στους τρεις, στα τρία λεπτά. Αρχίζουμε με τον κύριο Γκρό, συντονιστή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα και την παρουσίαση του προγράμματο τη Προεδρία σα. Καταρχά, βέβαια, σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία κατά την εκκίνηση κατά την των εργασιών σα με μειωμένη πρέπει να πω διάρκεια θητείας γιατί είχαμε και τώρα ένα μήνα των διακοπών και την καθυστέρηση που προκαλούν οι ευρωεκλογέ και την αναμονή του διορισμού της νέας ανάληψης καθηκόντων της νέας επιτροπής και άρα ασφαλώς έχετε πολύ μεγαλύτερη πίεση χρόνου και ξέρετε πολύ καλά ότι καμία προεδρία δεν μπορεί να ε, επαναπάβεται και να χάνει χρόνο. Τα θέματα τα οποία μας παρουσιάσατε είναι πάρα πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα η ασφάλεια ITS και μια και είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος μας θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω μια έλλειψη που παρατηρώ, ε, γενική έλλειψη, ότι δεν βρίσκω αρκετά φιλόδοξο το πρόγραμμά σας, ότι δεν έχετε πολλές ε, προσδοκίες εκφράσει, δεν διεκδικείτε δηλαδή, δεν έχετε πολλές φιλοδοξίες και Σα διαβεβαιώ εγώ ότι αν το πράτατε αυτό θα σε είχατε πάντοτε στο πλευρό σα το Κοινοβούλιο γιατί πάντοτε το Κοινοβούλιο στηρίζει οποιαδήποτε προεδρία αποφασιστικά και φιλόδοξα ε, προτείνει σχέδια και ε, προτάσεις. Για την Ευρωβινιέτα είναι τεράστια σημασία για το περιβάλλον ζήτημα και πιστεύω ότι και για το, για το Συμβούλιο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τεράστια σημασία το να ε, προχωρήσουμε με ομοφωνία, ανεξαρτήτως του αν υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές, πρέπει να προχωρήσουμε, να μην χάσουμε άλλο χρόνο όμως και να μην καθυστερήσουμε αναπτύσσοντας νέες μελέτε. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχει εξετάσει και το Κοινοβούλιο και βέβαια τα κράτη μας έχουν προσφέρει εν προκειμένου πολλές ε, πληροφορίες. Γι' αυτό λέω αφήστε βέβαια να γίνουν και αυτές οι μελέτε, αλλά εξασφαλίστε δυνατόν ταχύτερη πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Επίσης, ένα άλλο πολύ δύσκολο ζήτημα δεδομένης και της οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε τώρα, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση και ψηφοφορία χθε με τον προϋπολογισμό δείχνει ότι υπάρχει η πρόθεση να σας στηρίξουμε εάν έχετε και εσείς τη διάθεση να κάνετε πιο φιλόδοξα βήματα στο τομέα των μεταφορών διότι δεν μπορεί ο πολίτης να θεωρήσει ότι είναι αξιόπιστο να γίνονται επενδύσεις ε, μάλλον να γίνεται λόγος για επενδύσεις, για πολυλειτουργικές μεταφορές, για ε, νέα τεχνολογία, πιο ασφαλείς μεταφορές, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντο και να μην διατίθεται τα κατάλληλα κονδύλια μέσα από το προπολογισμό όταν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ και στο τομέα αυτό μην χάνετε άλλο χρόνο. Περιμένουμε το κύτταρο δυνατό κάποια μηνύματα ότι προχωρείτε. Και σας ε, διαβεβαιώνω και πάλι για την υποστήριξή μας. Ε, βιωσιμότητα, ε, βιώσιμες μεταφορές, συνδυασμένες μεταφορές και πάλι και εδώ τα δικαιώματα των επιβατών έχουν τεράστια σημασία και αν, τα, ε, αν σας απασχολεί το θέμα αυτό, εάν το περιλάβετε στο πρόγραμμά σας θα δείτε ότι και ο πολίτης θα σας ακολουθήσει, θα πιστεί για την επιλογή σα, για την ορθότητα τη επιλογή αυτή. Λυπούμε που δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερη συζήτηση στο θέμα αυτό στην Επιτροπή μα, γιατί θεωρώ ότι το μέσο των μεταφορών έχει τεράστιο ε, ρόλο να δραματίσει εδώ στην υπόθεση αυτή και όχι μόνο οι συνθήκε εργασία. Και νομίζω ότι ίσω θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ βεβαίω των αυτοαπασχολουμένων και του χρόνου εργασία, αλλά να μιλήσουμε και εμεί για τον ασφαλή χρόνο εργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφή νομοθεσία και σαφή μηνύματα για το χρόνο ανάπαυσης ξεκούραση του οδηγού και να μην μιλούμε μόνο για τι κοινωνικέ συνθήκε, γιατί δεν είναι μόνο η διάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων αυτών αλλά και η διάσταση τη ασφάλεια των μεταφορών εφόσον δεν διατηρείται επαρκή χρόνο ανάπαυση. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα και περιμένω πολύ καλή συνεργασία και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριο Σαλκαντράουι. Εσέντε. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την παρουσία της εδώ. Ομολογώντας ότι δεν φθονώ καθόλου τη θέση στην οποία βρίσκεται, διότι είναι πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο να λαμβεί κανεί ε, την προεδρία στις μεταφορές στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως είπε και ο κύριος Γκρός νωρίτερα, με νέο κοινοβούλιο, με νέα επιτροπή, με νέα συνθήκη πολύ σύντομα, αλλά και το αλλά είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, ε, δεν θα πρέπει αυτή η συγκυρία να ε, φέρει σε δεύτερο ρόλο ή να μειώσει τη σημασία των δραστηριοτήτων σας. Εδώ θα υπογραμμίσω ιδιαίτερα τη σημασία των θεμάτων που έχουν προχωρήσει και έχουν ήδη ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση σε επίπεδο κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα για, τις, για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών και τις βιώσιμες μεταφορές που έχουν τεράστια σημασία για την δική μου πολιτική ομάδα. Δεν άκουσα να γίνεται λόγος από την παρουσία σας ε, κυρία Υπουργέ για την έκθεση της κυρίας Αγέλα Σάντερε παραδείγμα για τις διασυνοριακές ή υπερσυνοριακές μεταφορές ή επί για την ε, δίωξη παραβάσεων ε, τον τομέα των υπερσυνοριακών μεταφορών. Πώς σκοπεύετε εσεί αυτή την ατιμορρησία η οποία επικρατεί ω προς τις διάφορες ε, παραβάσεις, παραβιάσεις ε, ε, στον τομέα αυτών να δράσετε. Μας λέτε ότι υπάρχουν 40.000 νεκροί το χρόνο. Ναι, αλλά αυτές, αυτοί οι θάνατοι, αυτές οι ζωές που χάνονται, χάνονται επειδή υπάρχουν αυτέ οι παραβάσεις από τον κωδικό, των κωδίκων οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, στην Ευρωβινιέτα Πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας ότι ε, έχει μεγάλη σημασία κλιματολογική ε, η διάσκεψη της Κοπενχάγης θα την αναλύσει την κλιματολογική αυτή σημασία και δεν μπορούμε να τη δούμε βέβαια αποκομμένη από το τομέα των οδικών μεταφορών. Αλλά πρέπει δυστυχώς να σημειώσω ότι αν δεν αποτολμήσουμε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, να κάνουμε κάποιες επιλογές, ε, πολιτικές επιλογές σημειώνω, δεν θα έχουμε επιτελέσει το έργο μας. Δεν θα έχουμε κάνει αυτό το οποίο καλούμεθα να πράξουμε. Επίσης, η εξωτερήκευση των, του ιστορικού κόστου των μεταφορών. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι θέλετε να μιλήσετε για το θέμα αυτό για το 2010, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο φάκελο που ήδη έχει συζητηθεί μια συζήτηση η οποία στρέφεται προς το μέλλον, ορίζει το μέλλον και νομίζω ότι πια πρέπει από τα λόγια να περάσουμε στα έργα. Η ομάδα μου λυπάται που η ε, Προεδρία δεν είναι σε θέση να προχωρήσει περισσότερο στο τομέα αυτόν. Θα υποχρεωθούμε λοιπόν να κάνουμε πολύ περισσότερα από το να θέσουμε μόνο το, να υπογραμμίσουμε το θέμα της τεχνολογίας και μόνο. Το ερώτημα λοιπόν αυτή τη στιγμή που τίθεται, μήπως εσείς μπορείτε να μας στείλετε μια, ένα θετικό και περισσότερο θετικό σήμα. Και βεβαίως ό,τι μας αποστείλει, το ντοσιέ που θα μας στείλετε, θα είμαστε επικριτικοί, ιδιαίτερα όσον αφορά την χρηματοδότηση για τα θέματα ασφαλείας των αεροδρομίων. Πιστεύω πως πάρα πολύ συγκεκριμένα θα μπορέσετε να εργαστείτε επί των φακέλων αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στέουξ από τους Φιλελευθέρους, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Φρονώ πως εδώ θα πρέπει να εργαστούμε κατά κάποιο τρόπο ούτως ώστε να εργαζόμεθα πάνω στους φακέλους του οποίου έχουμε αναχείρες και να μην ε, επηρεαζόμαστε από εξωτερικά γεγονότα τα οποία μπορούν να είναι επιβλαβή στην εργασία την οποία επιτελούμε. Αυτό που με ικανοποίησε από αυτά που είπατε, ότι υπογραμμίσατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα νεοποιημένο σύστημα μεταφορών. Σε, έχουμε μια εσωτερική αγορά ενιαία. Αυτό αληθεύει, ούτε, ούτε όντω ισχύει. Έτσι λοιπόν ο στόχος που έχετε θέσει είναι αρκετά δύσκολος και για μας ιδιαίτερα και οφείλεται αυτό στο Συμβούλιο καθότι το Συμβούλιο απαιτεί ομοφωνία και τέτοιου είδους πράξεις. Βλέπουμε αφετέρου πως έχουμε πάρα πολύ κόσμο τον οποίο θα πρέπει να πείσουμε και μεταπίσουμε όσον αφορά το θέμα αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι υπογραμμίσατε για την ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι κάτι για το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ καθώς επίσης ζητήσατε την απλοποίηση των διαδικασιών όσον αφορά την αυσιπλοεία. Κυρία μου πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι από αυτού του θέματος εισηγητής δηλαδή είναι οι μεταφορές οι διαθαλάσσεις σε όλη την ΕΕ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή μεταφορές οι οποίες δεν θα έχουν σκοπέλους οι οποίοι θα εμποδίζουν τη μετακίνηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε και λέγω ότι η μικρή, η παράκτια, η, η, η μεταφορά όταν είναι αναγκαία η χρήση της θαλάσσης για να μπορεί να γίνει κάλλιστα μία μεταφορά και δασυνοριακή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κυρία Πρόεδρε, είναι μία από τις προτεραιότητες αυτό το θέμα το οποίο σας θέλουμε. Και ξέρετε πράγμα πολύ καλά πως στην πρώτη ανάγνωση στείλαμε μία έκθεση του θέματος αυτού. Δυστυχώς η συνάδελφός μου η οποία είναι συντάκτη αυτό το θέμα δεν είναι εδώ παρούσα. Ωστόσο θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Κατά πόσο το Συμβούλιο φρονεί, κρίνει πως έχουμε ανάγκη όχι μόνο ε, συντονισμού αλλά και νομοθεσία αυτού του θέματο. Διαρωτάμε κατά πόσο πραγματικά θα πρέπει να νομοθετήσουμε επί του θέματο αυτού, ούτω ώστε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία επί των θεμάτων αυτών. Και εφόσον εμεί περατώσαμε την πρώτη ανάγνωση αυτού του θέματο, φρονείται αυτή τη στιγμή πω μπορεί κατά τη διάρκεια τη δική προεδρία να υπάρχει μια κοινή θέση επί των θεμάτων αυτών. Πράγμα το οποίο υπογράμμισε ο συνάδελφό μου προηγουμένω και, και το οποίο όντω είναι κάτι σημαντικό. Είναι μια απόφαση πολιτική ενεσχάτη στην αρχή των, των περιπτώσεων. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο έχουμε αφενό του υπουργού και αφετέρου του υπουργού οικονομικών. Οι υπουργοί οικονομικών θέλουν μόνο την ευρωβινιέτα και α, τελεία και παύλα. Ενώ εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή με την Ευρωβινιέτα να χρηματοδοτήσουμε τα εξωτερικά κόστη. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εγώ θέτω ένα ερώτημα και το οποίο είναι πάρα πολύ σύντομο η ερώτηση. Περιμένουμε πραγματικά το τέταρτο πρόγραμμα δράση επί των παρακτήων μεταφορών και τι ναυσιπλοεία και πιστεύουμε πω η Κομισιόν, μάλλον η, η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να γίνει αμέσω και η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια ανακοίνωση επί των θεμάτων αυτών. Θα πρέπει να ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσον εμεί μπορείτε να προσανατολίσετε την Κομισιόν κατά αυτόν τον τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει μία, ε, μία επιτάχυνση και να υπάρχει μία στόχευση πολύ καλύτερα από ό,τι προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τον πρώτο κύριο. Ο κύριος Κρέμερ έχει το λόγο παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ πολύ την Υπουργό για την παρουσία της εδώ και την εισήγησή της εκ μέρους ομάδας μου. Μιλήσατε για το περιβάλλον. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι χωρίς τροποποίηση της κινητικότητας, του είδους κινητικότητας που έχουμε επιλέξει, ε, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Έχει κατά τεράστια ποσοστά ε, συμμετοχή εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα ο τρόπος των μεταφορών που έχουμε στην Ευρώπη και από το 99 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά 30% το σύνολο των εκπομπών. Και γι' αυτό το λόγο έχει τεράστια σημασία η Ευρωβινιέτα γιατί έχουμε πολύ άνισες συνθήκες ανταγωνισμού. Η πρότασή μας λοιπόν της Ευρωβινιέτας είναι πολύ ενδοτικού χαρακτήρα θα έλεγα, πάλι δηλαδή δεν εξασφαλίζει τον ε, ισότιμο ανταγωνισμό και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται άλλες μελέτες. Οι μελέτες υπάρχουν, άλλες μελέτες δεν χρειαζόμαστε και γι' αυτό παρακαλώ προχωρήστε στη λήψη αποφάσεως. Αυτό είναι που χρειάζεται πλέον. 70% επίσης των, επενδύσεων ε, πηγαίνουν στις οδικές μεταφορές, στην κατασκευή δρόμων και όχι στους σιδηροδρόμους. Δηλαδή σε αυτό το οποίο προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να θέλουμε να υποδείξουμε τι θα πράξετε εσείς, θα ήταν προτιμότερο να ορίσετε ένα όριο στις επενδύσεις αυτές. Επίσης, έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο να ε, τεθεί σε εφαρμογή οδηγία για τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Μέχρι τέλους του έτους πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αυτή, αυτή η νομοθεσία και γι' αυτό θέλω να μας πείτε ποια είναι τα κράτη που δεν συμφωνούν στην εφαρμογή της. Και Ακόμη και στα τρένα υψηλή ταχύτητα, ξέρω βέβαια ότι κάποια κράτη έχουν δυσκολίε. Ε, θα ήθελα όμω να δω η Σουηδία τι στάση έχει στην υπόθεση αυτή. Η ε, επίσης παλαιά εκείνη η σύμβαση περί άλπεων Ξέρω ότι η Σουηδία απέχει γεωγραφικά και χιλιομετρικά πολύ από τις Άλπες, αλλά μην τη λησμονείτε, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί μες στο εξάμεινο αυτό. Επίσης, τα monster trucks τα γιγαντιαία λεγόμενα φορτηγά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μα είπε η εκπρόσωπό σα σήμερα το πρωί ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μα ασχολήσει. Αλλά εάν μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα φορτηγά από τον δρόμο στο σιδηρόδρομο θα κερδίζαν πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται όμως γίνεται το αντίστροφο. Αυτά τα τεράστια φορτηγά αντί να ε, φορτώνονται στη σιδηροτροχιά έρχονται όλο και περισσότερο σε περισσότερο ρυθμό, στους δρόμους μας. Επίσης ε, μη λησμονούμε ότι υπάρχουν και στις ε, μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές ανοιχτής θάλασσας αλλά και στις μεταφορές των εσωτερικών ε, υδάτινων οδών τεράστιες επιπτώσεις και εκπομπές, εκπτώσεις για το περιβάλλον και εκπομπές. Θα ήθελα να δοθεί σημασία και στο θέμα αυτό και βεβαίως να εξασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τις ιδροδρομικές μεταφορές. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω για του αυτοκινητοδρόμου, αν σκοπεύετε να προτείνετε ένα ενιαίο ανώτατο όριο ταχύτητα, γιατί η Γερμανία είναι το μόνο κράτο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει όριο ταχύτητα στου αυτοκινητοδρόμου τη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο. Ευχαριστώ, κύριο Ζέλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Υπουργό για την ε, παρουσία της εδώ, τα λόγια της και τις προτεραιότητες που ορίζει την επιμελητία δηλαδή και το ITS. Εμένα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα δικαιώματα των επιβατών, λεωφορείων, σιδηροδρόμων ε, που θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι το Δεκέμβριο Επίσης, στην οδηγία για τον ε, χρόνο εργασίας των ε, εργαζομένων σε οδικές μεταφορές θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να προχωρήσει και να παρακολουθηθεί η εφαρμογή της οδηγίας αυτής διότι έχουμε νομίζω αρκετές ε, διαφορές περιφερειακού χαρακτήρα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να δειχθεί κατανόηση για να έχουμε καλύτερη εφαρμογή τη οδηγία. Για την Ευρωβινιέτα επίση αναμένω περισσότερο φιλόδοξη στάση και μεγαλύτερη πρόοδο σε επίπεδο Συμβουλίου ω προ την έγκριση και εφαρμογή του συστήματο αυτού. Ύστερα από τρία χρόνια θα έχουν επιτέλου τα κράτη-μέλη να ε, εισαγάγουν εξαιρέσει από την εφαρμογή της ε, Ευρωβινιέτας Μέχρι τώρα η κατάσταση που επικρατούσε δεν ήταν πολύ λογική. Τώρα για τη Βαλτική θάλασσα. Μιλήσατε για τις μεταφορές, τα συστήματα μεταφορών, μιλήσατε για τις ε, προτεραιότητες Σουηδικής Προεδρίας. Ρωτώ λοιπόν, η ε, στρατηγική για την ε, Βαλτική συμπεριλαμβάνει και μια πιο καθαρή Βαλτική θάλασσα. Σημαίνει και πρόοδο, εξέλιξη στον τομέα αυτών. Όταν μάλιστα από τα εννέα κράτη που βρέχονται από τη Βαλτική το ένα μόνο, η Ρωσία, είναι μη ευρωπαϊκό κράτος και δεν τηρεί τις ε, προδιαγραφές και την νομοθεσία. Η Σουηδία πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ε, ασχοληθεί όχι μόνο με την νομοθεσία αλλά με την γενικότερη επίλυση ζητημάτων των μεταφορών και του περιβάλλοντος στη Βαλτική Ένα άλλο ζήτημα είναι οι τεράστιες διαφορές ε, και τα προβλήματα κυρίως ε, ε, στις οδικές μεταφορές μεταξύ Ρωσίας και Λιθουανίας. Είχαμε τεράστιες καθυστερήσεις στους δρόμους μας λόγω των κακών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Λιθουανίας, λόγω κακών συνθήκων ή πολιτικής στις οδικές μεταφορές. Πράγμα το οποίο βεβαίως έχει οδηγήσει σε τεράστιες κοινωνικές εντάσεις και προβλήματα. Και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει πάλι και με την εξωτερική πολιτική. Στη Βολτική έχουμε ένα ρωσικό καράβι. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και ίσως δεν θέλετε να τοποθετηθείτε, αλλά υπάρχει ζήτημα πειρατείας εις βάρος λιθουινικών και εστονικών ε, καραβιών. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, ο κ. Κόχλιτσεκ για την ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες ερωτήσεις θέλω να θέσω. Για τις μεταφορές στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Ξέρω ότι ε, η Τσεχική Προεδρία έχει δώσει σημασία στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Εσείς δώσατε στην θαλάσσια ναυσιμπλοεία. Ε, σε ό,τι αφορά ωστόσο τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές δεν πετύχαμε πολλά πράγματα. Ε, μιλάμε για την χρήση πλωτών υδάτινων δρόμων, έλβας, δούναβης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τι θα κάνετε. Ε, δεύτερο θέμα, μεταφορές Θα προχωρήσετε στο ΣΕΣΑΡ. Θα υπάρξουν κονδύλια επαρκή για το ΣΕΣΑΡ. Ιδιαίτερα για το συντονισμό του εναέριου χώρου. Τι φιλοδοξίες έχετε εκεί. Ποιους στόχους έχετε. Άλλο θέμα. Κατάρτιση των πιλότων. Πρόσφατα τα αεροπορικά ατυχήματα των οποίων γίναμε μάρτυρες, φαίνεται ότι οι πιλότοι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι στο να ε, πλανάρουν όταν σταματήσουν οι ε, κινητήρες. Αυτό μπορεί να είναι και θέμα, της, και θέμα κατάρτισης. Τι προτίθεστε να κάνετε για να μπορέσουν να μάθουν τεχνικές πλαναρίσματος οι πιλότοι. Συμφωνία ανοιχτή ουρανή με τις Ηνωμένε Πολιτείε τώρα. Υπάρχει μια δεύτερη συμφωνία με τη χώρα αυτή, το Open Skies, πόσο θα, πότε θα προχωρήσει και τι θα περιέχει. Συνδρομικές μεταφορές, το, σύστερα, το σύστημα TMS, τι θα κάνετε με αυτό. Θα έπρεπε να ενοποιήσουμε τα στάνταρ ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 27 διαφορετικά τέτοια πρότυπα. Επίσης, οδικές μεταφορές. Θα πρέπει να βελτιώσουμε καλύτερα οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων. πολλά από τα διασυνοριακά ατυχήματα οφείλονται σε αυτούς και στην έλλειψη εμπειρίας τους. Το ίδιο αφορά και τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Άλλο θέμα. Οι υπηρεσίες. Θέλετε να αυξήσετε τον αριθμό αυτών των οργανισμών ή να συγχωνεύσετε ορισμένε. Και επίσης, τι θα γίνει με τον Γαλιλαίο. Ευχαριστώ κύριε Κόλτσεκ. Σας δώσαμε δύο-τρεις ερωτήσεις κύριε Υπουργέ. Αν θέλετε να απαντήσετε σε έναν πρώτο γύρο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για τις πάρα πολύ σημαντικές ερωτήσεις τις οποίες υπέβαλαν. Ευχαριστώ επίσης για τη δέσμευση την οποία αναμβάνεται για την εξέταση αυτών των θεμάτων. Αφαιρθήκατε τις δυσκολίες που θα έχει αυτό το φθινόπωρο η Προεδρία μας. Μας, είπατε και μας κατηγορήσατε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στόχους και φιλοδοξίες. Ωστόσο έχουμε και τις δυσκολίες που ο Κύριο Κρόσ, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κατανόηση. Πρέπει να, είμαστε, να έχουμε κατανόηση. Κύριε Κρός, ο κύριος Ελκατροή και εσείς αναφερθήκατε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται ακριβώς αυτές οι φιλοδοξίες που έχουμε θέσει. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ όμως και στις δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε φέτος το φθινόπωρο. Ξέρετε ότι έχουμε ψηλά, ψηλές προδιαγραφές, ψηλούς στόχους και θα θέλαμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους όσον αφορά τις μεταφορές. Αλλά θα πρέπει να εμβαθύνουμε τα θέματα αυτά και πρέπει να βαθύνουμε ακριβώ διότι έχουμε αυτέ τι ψηλέ προσδοκίε και θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά του τομεί καθώ επίση και τι εργασίε οι οποίε θα πρέπει να γίνουν για την κατάτμιση και κατανομή αυτών των, εργασιών και το πώ θα πρέπει να γίνουν. Ευελπιστώ πω τα δύο αυτά κοινοτικά όργανα θα εργαστούν επιμελώς για να υπάρχουν απτά καλά αποτελέσματα αποδεκτά από τους πάντες. Ξέρετε πως έχετε μεταφορές οι οποίες θα είναι μόνιμες, αϊφόρες επίσης. Ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται πάλι και πολλά και αυτός είναι και ο, ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος με μά αυτή τη στιγμή αναφερόμενο σε αυτό το θέμα και εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να συμμετέχετε κι εσείς ως βουλευτές σε αυτές τις δραστηριότητες που αναφέρω. Προφανώς Όλα αυτά γίνονται ενώπιον δύο προκλήσεων τις οποίες έχουμε. Καταρχήν υπάρχει παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυτή η κρίση μας υποχρεώνει να θέσουμε ορισμένους στόχους και φιλοδοξίες, ιδιαίτερα πριν από την συνάντηση της κορυφής της Κοπενχάγης. Θα θέλαμε να, να προωθήσουμε την οικονομία αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια προστασία της οικολογίας, να λεφθεί υπόψη η οικολογία και αυτό θα πρέπει να γίνει εκ μέρους όλων των παραγόντων κύριο που συμμετέχουν. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια ομοιομορφία στον τομέα των μεταφορών. Αυτό έχει σχέση και την απασχόληση, αλλά έχει μια αρνητική επίπτωση όσον αφορά τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την επιβίωση. Κύριε Γκρός, αναφερθήκατε στο θέμα των δικαιωμάτων των ε, επιβατών του δικαιώματος του πολίτη. Επιμείνει σε αυτά τα θέματα. Ο πρόεδρος μας επίσης επιμένει από αυτού του σημείου. Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης και κινητικότητα των πολιτών μας. Ωστόσο αυτό πρέπει να ειδωθεί μέσα στο ένα πλαίσιο της καταστάσεως της παρούσας των μεταφορών μια ετερογένεια και ετερομορφία η οποία υπάρχει μεταξύ των διαφορών χωρών και θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των εταιριών, επιχειρήσεων και των πολιτών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί. Κύριε Ελκατραουή, αναφερθήκατε σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ειδικό, δηλαδή όσον αφορά εκείνα τα εγκλήματα, και τα δικήματα καλύτερα, τα οποία γίνεται διασυνοριακά και κατά πόσο πραγματικά αυτή τη στιγμή τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες σε αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή και να καταλάβουμε, όπως το έλεγε και προηγουμένως, ότι εμείς ε, πραγματικά υπογραμμίζουμε το θέμα της ασφάλειας πολύ περισσότερο στα πλαίσια της ΕΕ. Με τη σειρά του θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα νομικό εργαλείο, αλλά βεβαίως έχουμε και ένα πρόβλημα νομικής βάσης όσον αφορά το θέμα αυτό. Ίσως η συνθήκη της Λισαβόνος θα μπορέσει να μας βοηθήσει να επικουρήσει αυτό το θέμα. Αλλά όσον αφορά αυτό το θέμα θα πρέπει κύριε Κατρογουή να σας διαβεβαιώσω πως έχουμε μεγάλους στόχους, μεγάλες ε, προσδοκίες και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βρούμε και τομική βάση ούτως ώστε να υλοποιήσουμε αυτά τα, αυτές τις προσδοκίες. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωβινιέτα, ξέρω είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ε, ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί εξημών το έχουν αναφέρει ο κ. Κράμερ, δεικτικά λέγω το όνομά του, αλλά και άλλοι. Ο κ. Κόλιτσεκ, Στέρξ, όλοι αναφέρθησαν σε αυτό το θέμα της Ευρωβινιέτας. Μια μια εισέτη φορά θα ήθελα να επαναλάβω πως και εμείς θα θέλαμε πραγματικά να έχουμε αυτά αποτελέσματα σαν Προεδρία. Πλην όμως πολλά κρατημέλη ε, παραμένουν σκεπτικιστές όσον αφορά το κόστος και τη χρησιμότητα της Ευρωβινιέτας. Κατά πόσο πραγματικά τα προσδοκόμενα αποτελέσματα θα είναι αυτά που πραγματικά θέλουμε κατά πόσον θα μειώσουν ε, ε, την επίπτωση που έχουν οι μεταφορές όσον αφορά το, το κλίμα, την κλιματική αλλαγή. Ε, όπως το έλεγα προηγουμένως, θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε σοβαρά τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε αναχείρες και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή έχει σχέδια να κάνει μία ε, προσωμείωση όσον αφορά τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα με τα στοιχεία τα οποία μας υπευλήθησαν εκ μέρους των κρατών μελών ενδεικτικά θα λέγαμε όσον αφορά την Ευρωβινιέτ. Από τη στιγμή εκείνη η οποία η Κομισιόν θα επανέλθει με μελέτες και με στοιχεία και με τεκμηρίωση, εμείς θα αναλάβουμε πλήρως στα πλαίσια του Συμβουλίου αυτό το θέμα και θα το θέσουμε εκ νέου. Νομίζω πως θέλετε αυτή τη στιγμή να έχετε μια απάντηση η οποία θα καλύπτει όλους τους τομείς, τους τομείς όσον αφορά την Ευρωμηνιέτα. Ωστόσο θα πρέπει τα αποτελέσματα να είναι απτά, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και συμφωνώ με τον κύριο Καβέλιο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να διαθέτουμε μια ικανότητα σιδηροδρομική τέτοια η οποία θα μας επιτρέπει να γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές και μεταφορές μέσω του, των σιδηροδρόμων. Ασφαλώς είναι ένας στόχος αυτός, φιλόδοξος, είναι μια ευχή αν θέλετε. Αλλά συνειδητοποιώ αφετέρου πως αποτελεί θέμα ευρωπαϊκής συζήτησης. Ποια είναι εκείνα τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να φτάσουμε να έχουμε ένα πιο αποτελε... μια πιο αποτελεσματική μεταφορά διακρατική για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις κλιματολογικές που έχουμε ενώπιόν μας. Ο κύριος Κρέμερ αναφέρθηκε επίσης σε αυτό το θέμα. Ο τομέας των μεταφορών έχει ένα ρόλο και μια εντολή. Αληθεύει αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως όσον αφορά τις, ποσός, τις που υπάρχει για τη συνολική ρήπανση η οποία δημιουργεί Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αναφερόμαστε συνεχώς αυτά τα θέματα όσον αφορά τη, την συμφωνία της και την σύγκληση της Κοπενχάγης μόνο για τις αυξήσεις της συνεργασίας με το Καρτόν μελών όσον αφορά των μεταφορών τότε θα δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή εκείνα τα στοιχεία, εκείνες οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να κατανείμουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα και να ανοίξουμε αυτή τη νέα λεωφόρο εντό εισαγωγικών για βελτίωση των πραγμάτων στο μέλλον. Ειδικότερα θα αναφερθώ τώρα στο θέμα για τον φορτηγών, των πολύ μεγάλων φορτηγών. Όντω έχουμε στη Σουηδία μια εμπειρία επί ε, αυτών των φορτηγών. Δεν θα θέλαμε όμω ουδαμό και οι υπόλοιπε χώρε να ακολουθήσουν το δικό μα παράδειγμα υποχρεωτικά. Εν πάση περιπτώσει, φρονώ πω εάν ενδιαφέρεστε, εγώ μπορώ να σας καλέσω να δείτε πραγματικά πώς λειτουργεί το δικό μας ε, σύστημα επιτόπου να το δείτε και να δείτε πραγματικά ποιες είναι οι επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος από αυτά τα υπερφορτηγά. Διότι μειώνει τον αριθμό των φορτηγών στους οδικού, στην οδική μεταφορά. Επίσης το θέμα των Άλπαιων είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι διακρατική και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτή τη Επιτροπή και εφόσον τελειώσουν οι εργασίε τη, πραγματικά θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Τότε αναφορά τώρα τη στρατηγική της, Βαλτική, Βαλτικής, συγγνώμη, την οποία αναφέρει ένας άλλος συνάδελφος, οφείλω να πω πως αυτό το οποίο είπατε πραγματικά κύριε Ζήλε είναι μέσα στους στόχους της Σουηδικής Προεδρίας. Βεβαίω, η βαλτική στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική, η αποτελεσματικότητα αυτών των μεταφορών στη βαλτική είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίω ε, η στρατηγική της βαλτικής έχει τον ρόλο τον οποίο θα πρέπει να παίξει σε αυτά τα πλαίσια. Θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν διάδρομοι Ανατολής, Δύσης, Δύσης, Ανατολής οι οποίοι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί αυτοί οι διάδρομοι και να υπάρξει μια ομοιογένεια και μια ενότητα στα πλαίσια της ΕΕ Ανατολής Δύσης. Τόσο όσον αφορά συγγνώμη αυτά που είπε ο κύριος Κολιτσέκ για το Σεζάρ, οφείλω να ομολογήσω πως παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη του, της διαδικασίας όλης αυτής. Είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση της εξέλιξης Στη συνέχεια και τη ανάπτυξη Στη συνέχεια το Συμβούλιο θα μπορεί να δράσει πολύ πιο άμεσα εφόσον αυτές όλες οι πέρα το περατωθούν. Την επίδραση τώρα της αερο των αερομεταφορών επί του περιβάλλοντος. Έχουμε πάρα πολύ καλές εμπειρίες προσεγγίσεις με πλανάρισμα οι οποίες είναι πάρα πολύ πιο οικολογικές, ε, ε, οι οποίες αποφεύγουν την κατανάλωση πάρα πολύ κα, ε, κατανάλωσης καυσίμων. Στο ΣΕΖΑΡ βεβαίως θα υπάρξει μια δυνατότητα καλύτερη εφαρμογή αυτών των, αυτών των σχεδίων, των project και όσον αφορά την διαπραγμάτευση μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης τον Οκτώβριο θα γίνει και ευελπιστούμε πως πραγματικά θα υπάρξει πρόοδος με τους Αμερικανούς πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τούδε. Τώρα, όσον αφορά τις εσωτερικές ναυσιπλοίες και τους ε, Η Τσεχική Προεδρία, η οποία άνοιξε πρώτη αυτή την υπόθεση, ε, θέλει η Σουηδική Προεδρία να ακολουθήσει αυτή τη συζήτηση η οποία προϋπάρχει αλλά προς το παρόν δεν έχουμε φακέλους, δοκουμέντα τα οποία όσον αφορά τις εσωτερικές ε, με, ε, μεταφορές Εκτός από τα δικαιώματα των επιβατών και τη συμμετοχή των οδών αυτών, των καναλιών αυτών, τα οποία αφαιρεθήκατε στις προηγούμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω 7 μέλη αυτή τη στιγμή. Εάν παραμείνουμε πραγματικά στο χρονοδιάγραμμα θα παρακαλούσα τα μέλη να μείνουμε σε δύο λεπτά μόνο εφόσον έχουμε την Υπουργό αυτή τη στιγμή και να μπορέσει να έχει πέντε λεπτά. Η κυρία Ντιβεράκη είναι πρώτη για να μπορέσει και η Υπουργό να απαντήσει παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που στενοποιώ μα για να μα παρουσιάσει το πρόγραμμα τη Σουηδική Προεδρία. Τρει ερωτήσει στι αερομεταφορέ. Πρώτον, αφορά τη χρηματοδότηση όσον αφορά την ασφάλεια. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σαφέ ότι το χρηματοδότηση αυτό δεν θα πρέπει να είναι ει βάρο των επιβατών και τα κράτη πρέπει να χρηματοδοτήσει. Κατά πόσο η Σουηδική Προεδρία φρονεί πω μπορεί να έχει μια κοινή θέση επί θέματο αυτό μέχρι το τέλο τη χρονιά. Δεύτερο, έχει σχέση με την ασφάλεια των αερομεταφορών. Ξέρετε, του τελευταίου μήνε είχαμε μεγάλε. Ε, πολλά ατυχήματα μάλλον και η Κομισιόν ετοιμάζει ένα κείμενο όσον αφορά την πτώση αυτών των αεροπλάνων και το οποίο θα προσιαστεί τον, το φθινόπωρο. Κατά πρώτο, η Προεδρία πρόβλεψε να δώσει μία προτεραιότητα σε αυτό το κείμενο που θα έρθει από την Κομισιόν. Τρίτη ερώτηση και παρακολουθήσαμε του σύνεγγυ την οδηγία όσον αφορά το σύστημα EDS ε στο οποίο θα υπήρχε το σύστημα της αερομεταφορών στο οποίο προέβλεπε όλε εκείνε οι τοπίε που έρχονται στην Ευρώπη θα πρέπει να ελέγχονται, ούτω ώστε να μην υπάρχουν κυρώσει μόνο εναντίον μια εταιρεία και να υπάρχει στρέβλωση τη του ανταγωνισμού. Κατά πόσο στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση αυτή τη στιγμή θα προτείνει κάτι τέτοιο, ώστε να υπάρχει διεύρυνση του ευρωπαϊκού σύστηματο σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υπάρξει μια καλύτερη κατανομή κατά αυτόν τον τρόπο, ούτω ώστε οι αερο οι να μπορούν αυτή τη στιγμή ε, να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή αλλά χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φέρει όλα τα άχθη αυτής της προσπάθειας η οποία αναπτύσσεται. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η επόμενη ομιλήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Ο κύριος Αρκατρουή, ο συνάδελφος... Α, εδώ, εδώ είμαι κυρία μου, κύριε Υπουργέ, εδώ είμαι, μπροστά σας. Ο συνάδελφό μου λοιπόν, ο κ. Σαρκατρούη, ανέφερε ένα θέμα και, και ε, καταλαβαίνω ότι είστε κουρασμένοι κύριε Υπουργέ. Είναι η συγγήτρια Υπουργέ, όσον αφορά τις κυρώσει που θα πρέπει να ε, επιβληθούν διασυνοριακά. Αυτή την έκθεση έχω. Η χώρα σας είναι εκείνη η οποία παρουσίασε πολλές, πολλά πολλέ αντιρρήσει όσον αφορά την νομική βόση, αλλά η Σουηδία φαίνεται, ενδιαφέρεται πάρα πολύ όσον αφορά την ασφάλεια και εμείς θα είμαστε λίγο πιστευτοί αν πούμε πως είμαστε υπέρ τη μειώσεως της ταχύτητας και των θυμάτων αλλά όταν υπάρχει ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θέλουμε να εφαρμοστεί όσον αφορά αυτά τα δικήματα τα οποία διαπράττονται και έχουν σχέση με όλα τα κράτη-μέλη, τα 27 ενώ, και βλέπουμε σε αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μία από τι λίγε χώρε οι οποίε αντιστέκεται σε αυτό το σχέδιο. Διαρωτώμε κατά πόσο το Συμβούλιο θα βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει ένα ξεμπλοκάρισμα όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Μετά τις εκλογές που είχαμε πρόσφατα, νομίζω πως πραγματικά οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις μεταφορές, ιδιαίτερα στα Κέντρο των πόλεων. Η Στοκόλμη αποτελεί εξάλλου ένα παράδειγμα σε αυτό το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη διάρκεια, συμφωνώ με το συνόδευμα, με τον συνάδελφο Κατρογουή, όσον αφορά και τη βινιέτα, Ευρωβινιέτα, έχουμε ανάγκη αυτή την Ευρωβινιέτα, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο της κρίσης, αλλά οι πολίτες θέλουν περισσότερη σιγουριά. Ας και ιδιαίτερα στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια προβλήματα όσον αφορά με τους σιδηροδρόμους καθώς επίσης και με τους ε, θαλάσσιους υδάτινους αυτοκινητόδρομους θα έλεγα, οδούς. Το Κοινοβούλιο τώρα αυτή τη στιγμή θα ήθελε αυτή να υπάρξει μία αποκατάσταση ενός συστήματος και επέμεινε πάρα πολύ καλά όσον αφορά αυτά τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσο η Σουηδική Προεδρία θα υποστηρίξει αυτό το αίτημα το οποίο υπάρχει και όσον αφορά τη διάρκεια θα πρέπει και το διαρκή χαρακτήρα θα πρέπει να συζητήσουμε για την αποτελεσματικότητα τη λογισμική, όχι μόνο την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, καθότι η Σουηδία έχει πολλές επιχειρήσεις όπως η IKEA, το IKEA το οποίο στρέφεται πολύ περισσότερο προς το σιδηρόδρομο και ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουμε μια καμπάνια πώς πραγματικά τα εμπορεύματα αυτά έρχονται μέχρι το σπίτι τους και μέχρι τη χώρα τους. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν αφορά ε, το, τις μεταφορές. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. Προσβλέπουμε ω Επιτροπή Μεταφορών στη συνεργασία με την Προεδρία. Ε, θα συμφωνήσω με τον ε, κύριο Κόξ ότι θα επιθυμούσαμε ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά ξέρω και αντιλαμβάνομαι τι δυσκολίε που υπάρχουν ε, αυτή την περίοδο. Με ικανοποίηση άκουσα την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην ασφάλεια των μεταφορών και ιδιαίτερα των αερομεταφορών και ε, ειλικρινά λυπάμαι που αισθάνομαι σήμερα την υποχρέωση και το καθήκον να ενημερώσω και εσάς αλλά και την Επιτροπή Μεταφορών για ένα ε, δυσάρεστο ε, συμβάν των τελευταίων ημερών. προχθές, την 31η Αυγούστου, κυρία Υπουργέ, οι επιβάτες της πτήσεως 983 των Ολυμπιακών Αερογραμμών που πετούσε εντός εθνικού εναερίου χώρου κράτους μέλους, δηλαδή της Ελλάδας, κυριολεκτικά έντρομοι για την ασφάλειά τους είδαν από τα παράθυρα του αεροσκάφους τους σε απόσταση 100 ποδών, δηλαδή 30 μέτρων, ένα τουρκικό πολεμικό αεροσκάφος τύπου F-16 να παρενοχλεί την πτήση τους. Το σοβαρό αυτό συμβάν δεν είναι μεμονωμένο και έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της επίμονης τουρκικής πολιτικής μιας υποψήφιας χώρας να μην υποβάλλονται σχέδια πτήσεων από τα στρατιωτικά της αεροσκάφη όταν μπαίνουν στο Flight Information Region της, ε, των Αθηνών. Τα όρια αυτής της περιοχής έχουν καθοριστεί από τον ΑΙΚΑΟ. Το ζήτημα δεν είναι ούτε ελληνοτουρκικό, ούτε στενά πολιτικό. Αφορά την ασφάλεια των πτήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ασφάλεια των αερομεταφορών ήταν ανέκαθεν και ευτυχώς μία από τις πιο κρίσιμες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτής της Επιτροπής, της Επιτροπής Μεταφορών. Θέτω λοιπόν το σοβαρό αυτό ζήτημα υπόψη σας κυρία Υπουργέ και μέσω ημών στο Συμβούλιο ε, προκειμένου να το θέσετε κι εσείς στις επαφές σας με τους Τούρκους αξιωματούχους. Το θέτω υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται εκπρόσωπός της εδώ εν ώψη της σύνταξης της έκθεσης προόδου για την Τουρκία που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο και βεβαίω το θέτω για να καταγραφεί υπόψη της Επιτροπής Μεταφορών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαντέλεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ακούσω τη δική σας απάντηση, αντίδραση όσον αφορά την εναρμόνιση των απαγορεύσεων, όσον αφορά την οδήγησε στην Ευρώπη. Νομίζω πως είναι απλές αυτό που πραγματικά συνάδει με τους στόχους της Σουηδικής Προεδρίας. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις όσον αφορά τα, διακίνηση των φορτηγών στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει ένα πλάνο όσον αφορά τις ώρες οδήγησης στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι υπάρχουν πάρα, πολλέ, ε, πάρα πολλά χιλιόμετρα τα οποία γίνεται επιπλέον καθώς επίσης και μια περιττέρω μόλυνση του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να επιμείνετε επιτραφέντε αυτό το θέμα πώς ακριβώς θα πρέπει να γίνει η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Η Γερμανία, για παράδειγμα, απαγορεύει την Κυριακή. Είναι, ο βασικός, είναι η βασική χώρα που η κυκλοφορία γίνεται και οι μεταφορές γίνονται διαφορετικών και αυτό στο σύνολο των Ευρωπα... της Ευρώπης έχει αυτή όμως τη θέση η οποία είναι πάρα πολύ βασική και κεντρική για την εναρμόνιση δηλαδή επαναλαμβάνω ότι δεν θα κυκλοφορούν τα φορτηγά της, την Κυριακή. Εγώ είμαι υπέρ τη αρχεία τη Κυριακή. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν να πάνε στην εκκλησία θέλουν. Αλλά θα ήθελα πραγματικά τη συγκεκριμένη σα θέση όσον αφορά αυτή την απαγόρευση κυκλοφορία τη Κυριακές. Κατά πόσον επίσης θα ήθελα να ξέρω η Ευρωβινιέτα να έχει σαν στόχο να γίνει μια μεταφορά από τις οδικές μεταφορές προς το σιδηρόδρομο. Όχι μόνο προς το ΡΑΙ, αλλά προς το σιδηρόδρομο, αλλά και προς άλλους ε, πάλι μεταφορές. Θα ήθελα να το πείτε πολύ σαφώς. Ο κύριος Κοκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θεωρώ... Ναι, εδώ στο, κέντρο. Βλέπω ότι έχετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, διότι σημαντικό για μένα δεν είναι το πόσα προγράμματα, το πόσα σχέδια θα προτείνετε, αλλά το τι ποιότητα θα είναι αυτά. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα θέλω να αφαιρθώ, παρακαλώ, στο e-call το ηλεκτρονικό σύστημα ε, τηλεφωνημάτων έκτακτης ανάγκης να βοηθήσετε να προχωρήσει η υπόθεση και επίσης δεδομένου ότι η Επιτροπή μας είναι η Επιτροπή των Μεταφορών και του Τουρισμού θα ήθελα να σημειώσω ότι ο τουρισμός είναι άριστο μέσο για να οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που είστε μεταξύ μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπες μέχρι τούδε. Ο λόγος υπήρξε έκτακτος, καταπληκτικός, ωστόσο επιτρέψαμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις ότι και αυτό είναι και το ότι ήταν πάρα πολύ γενικό ο λόγος αυτό βέβαια, τα θέματα είναι πάρα πολύ περιπλοκό, πλην όμως το σύστημα της ε, Προεδρίας είναι ένα σύστημα μεταλαμπάδευσης της Προεδρίας από χώρα σε χώρα, αυτός είναι θα σας ζητήσω ασπαζόμενος αφενός τα λόγια τα οποία είπατε προηγουμένως θα σας ζητήσω να ε, αυτά τα οποία είπατε να έχουν να άπτονται του της κοινή λογικής διότι Ξεκινάω από το θέμα της Ευρωβινιέτας. Ξέρετε ότι πρόκειται περί μεγάλης διαφοράς η οποία υπάρχει από χώρα σε χώρα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί και να μην κάνουμε μεγάλες άλματα και κενά όσον αφορά το μέλλον. Η διαφορά της Ισπανίας είναι πάρα πολύ γνωστές ποιες είναι αυτές οι διαφορές και έχουμε διαφορετικά κριτήρια όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά κυρία Υπουργέ η πρώην Υπουργό ε, Μεταφορών της χώρας μου είναι εδώ και ασπάζεται ευελπιστό της απόψης μου. Δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε μεγάλες ε, περιπέτειες και να παραλείψουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω το έχει ερώτημα. Σε κατά πόσον η Σουηδική Προεδρία θα κατορθώσει να καταλήξουν σε εκείνες οι, διασ... οι προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από τις πρόεδρες προεδρίες και ποιες είναι οι δεσμεύσεις τις οποίες έχουν για να το κάνει και επί Ισπανικής προεδρία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρξει, υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ των δύο Προεδρίων, Ισπανικού και Σουηδικού και θα ήθελα να ξέρω πραγματικά ποια θα είναι αυτή η μεταλαμπάδευση η οποία θα γίνει μετά την ε, αναχώρηση της Σουηδικής Προεδρίας και θα, ξέρουμε, θα θέλαμε επίσης να θέσουμε να υπογραμμίσουμε μάλλον τα κείμενα εκείνα τα οποία άπτονται αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων. Θα ήθελα εκ περισσού να γνωρίζω ποιες είναι εκείνες οι προσπάθειες οποίες θα αναλάβετε σε σχέση με αυτές τις δυσκολίες ε, τα θέματα τα διασυνοριακά για να μπορούν να υπάρξουν και να λειτουργήσουν αυτά τα δίκτυα που ανέφερα. Ευχαριστώ. Κυρία Αλβαρέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσία στην οποία μας κάνατε. Ένα από τα στοιχεία τα οποία έχετε αναφέρει είναι πάρα πολύ σημαντικό ήδη Όπως το είπε ο κ. Γκράντες, εγώ υπήρξα υπουργό μεταφορών πριν από λίγο καιρό και γνωρίσαμε, συνέβη ένα τύχημα της Σπανέρ που ήταν πάρα πολύ σοβαρό Κατόπιν τούτου και άλλων ατυχημάτων διαπιστώσαμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να τροποποιηθεί η οδηγία όσον αφορά την έρευνα των ατυχημάτων και τις πληροφόρηση όσον αφορά τα ατυχήματα τα οποία γίνονται. Το βασικό στοιχείο αυτής της νομοθεσία έχει σχέση όσον αφορά με τα απορίσματα, συμπεράσματα των ερευνών που γίνονται και των ακρίσεων. Υπάρχει μια προκαταρτική η οποία γίνεται και η οποία έγινε από την Ισπανική ε, Επιτροπή Ελέγχου αλλά υπάρχει και μια διεθνής επιτροπή, εταιρεία, η οποία είναι αμερικανική και θα σας ζητήσω αυτή τη στιγμή, ναι, για αυτές τις συστάσεις που έχουν γίνει μέχρι τούδε θα πρέπει να καταλήξουν, διότι μετά από αυτό το ατύχημα ζητήσαμε εμεί όπως οι αρχές αυτές να θέσουν ε, στη διάθεση όλες αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν στους επιβάτες. Διότι αυτό απαιτεί όχι μόνο τον επιβατών αυτών καθευτών, αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία μπορεί να καταλήξει σε πολλές ε, μπορεί να γλυκάνει την ψυχή αν θέλετε πολλών ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει προσφυλή τους άτομα σε ατυχήματα, αεροπορικά ατυχήματα. Οι, οι οικογένειες λοιπόν των εκλειπώντων μπορούν να έχουν τέτοιου είδους πληροφόρηση η οποία θα τους καταπραίνει όπως είπα προηγουμένως επίσης θα μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια προσπάθεια όσον αφορά τη μαύρη λίστα για τις αεροπορικές εταιρείες Ξέρουμε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εργάζεται επί του θέματος αυτού θα πρέπει να γίνουν τάχοι να επιταχυνθεί για να μην υπάρχουν τέτοιου ατυχήματα στο μέλλον Ευχαριστώ πάρα πολύ Η κυρία Λίχτενμπεργκερ Πρόεδρε ευχαριστώ και θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις θα ήθελα να ρωτήσω εάν σκοπεύει η Υπουργό να ασχοληθεί με το θέμα των ε, δικαιωμάτων των επιβατών στην περίπτωση επεισοδίων όπως αυτής της ε, εταιρείας όχι Air Berlin, αλλά μια άλλη, δεν θυμάμαι το όνομά τη, που. Ε, Sky Europe, ναι, αυτήν που έκλεισε και ρίξε πτώχευση. Και οι επιβάτες μένουν μετέωροι χωρίς καμιά ελπίδα για αποζημίωση. Επίσης, για τα τεράστια φορτηγά, για τα υπερφορτηγά. Δεν νομίζω ότι είναι συνενετική η θέση που ακολουθείτε. και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Επιτροπή των Μεταφορών και στο παρελθόν, δηλαδή να, κάνει, να προβεί σε αξιολόγηση των κοινωνικών και πολιτικών δαπανών ή του κόστους που θα σήμαινε η μετατροπή των ε, σιδηροτροχιών ε, ώστε να προσαρμοστούν σε αυτά τα τεράστια φορτηγά, τα υπερφορτηγά. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην ερώτηση για την ε, σύμβαση των Άλπιων, στην οποία δεν έχετε δώσει απάντηση. Και επίσης το θέμα για την Ευρωβινιέτα. Σημειώνω επίση ότι το να κάνετε άλλε 15 μελέτε επιπτώσεων ε, δεν πρόκειται να συμβάλλει σε τίποτε. Μόνο να επιβαρύνει τη διαδικασία. Δεν πρόκειται να μα βοηθήσει να βρούμε λύση για δε τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας θα πρέπει να ε, προσφέρουμε το ελάχιστο πιστεύω σύνολο κοινών προδιαγραφών και όχι να επιδιώκουμε την εναρμόνιση. Γιατί πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με απαγορεύσεις που έχουν, να που έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή ε, απαγόρευση κυκλοφορίας στη νύχτα ή απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές ε, με υψηλό ποσοστό τουρισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας και το καθεξής. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω ικανοποιητικά. Ας ξεκινήσουμε με το ζήτημα της ασφάλειας των αέριων μεταφορών. Φυσικά θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό και στη διάρκεια της Προεδρίας μας όπως είπα και κατά την ε, παρουσίασή μου. Στο τομέα λοιπόν αυτών Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να, ε, γίνεται, να, να υποβληθεί η πρόταση και να εκδηθεί εγκαίρως, ώστε να ε, αντιμετωπιστεί σοβαρά και υπεύθυνα το ζήτημα της ασφάλειας των μεταφορών με τις διαδικασίες ε, και τις διατάξεις που θα ισχύουν σε περίπτωση ε, διερεύνησης ή ανάγκης διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων. Γενικά τώρα για τις ενέργειες μεταφορές. και τα δικαιώματα ανταλλαγή εκπομπών καυσαερίων. Έχουμε συμφωνήσει επί ενός συστήματος ανταλλαγών εκπομπών και στις γενικές συζητήσεις σκοπεύουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε και τα οικονομικά μέσα τα οποία έχει και στο παρελθόν μετέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο και ελπίδα να εξασφαλίσουμε ε, συμφωνία σε ένα συνολικό επίπεδο. Αλλά φυσικά θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία την οποία μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για, τα, ε, για τις υπερσυνοριακές παραβάσεις και τα σχετικά πρόστιμα που αναφέρει η κυρία Γιάλα Σάντερ. Πολλές είναι συζητήσεις ως προς την νομική βάση, όπως είπα και νωρίτερα, και πρέπει ασφαλώς να σεβαστούμε την ε, δεδομένη νομική βάση. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, όταν τεθεί σε εφαρμογή, εφόσον τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί αυτομάτως. Θα επιληθεί αυτομάτως. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω λέγοντας ότι όταν μιλούμε, όταν έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια των ε, μεταφορών, πάντοτε συμφωνούμε στον γενικό στόχο. Αλλά δυσκολίε αντιμετωπίζουμε όταν έρχεται η ώρα για συζήτηση τη νομική βάση συγκεκριμένα ή του πυλώνα στον οποίο θα υπαχθεί. Πάντως, με τη συνθήκη της Λισαβόνα, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα αυτομάτως αντιμετωπίζεται. Επίσης, η κυρία Γιάλα έθεσε μια ερώτηση ως προς τις ε, συνδυασμένες μεταφορές συνδυασμένες μεταφορές οι οποίες αποτελούν σαφώς προτεραιότητα για τη Σουηδική Προεδρία με στόχο τις πιο αποτελεσματικές ε, μεταφορές με ελάχιστο, ελάχιστες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και με όσο το δυνατόν πιο οικονομικό κόστος. Αυτός είναι ο στόχος μας. κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας θα γίνει διάσκεψη για τα ε, ΤΕΝ και τις ε, υπερσυνοριακές μεταφορές. Η κυρία Γιάλα επίσης αναφέρθηκε σε μια εταιρεία. Ναι, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι έχει τεράστια σημασία το να εμπλακεί και ο χώρος της οικονομίας των επιχειρήσεων, δηλαδή σε αυτές μας τις προσπάθειες, ώστε να απτυχθούν μεταφορές με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερες εκπομπές. θεωρώ ότι είναι θετικό το να καταβάλλονται προσπάθειες σε αυτό το στόχο. Και σύμφωνο με τις προτεραιότητες της Ειδικής Προεδρίας για το μέλλον των μεταφορών. Επικεντρωθήκαμε στην ε, συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ανάλυση της κατάστασης και της προτάσεις που θα για το μέλλον των μεταφορών κατά τη διάρκεια της Ουδικής Προεδρίας. Για τον κύριο Κουμουτσάκο. Αναφερθήκατε κι εσείς στην ασφάλεια των ε, επιβατών και για άλλη μια φορά θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι έχει τεράστια σημασία να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες γι' αυτό συνθήκες. Θα καταβάλω κάθε δυνατή ε, προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλύτερη πρόσβαση, καλύτερη κινητικότητα για τους πάντες. Για τον κύριο Βάλτερ. Αναφερθήκατε στην εναρμόνιση των απαγορεύσεων κυκλοφορίας. Ναι, πολλά από αυτά βέβαια θα πρέπει να κρίνονται σε επίπεδο εθνικό, κατά περίπτωση. Και όπως ήδη υπόθηκε υπάρχουν ε, ε, περιφερειακού χαρακτήρα διαφορές. Ε, είτε πρόκειται για το, την επιβάρυνση, τον, την εισφορά τη λεγόμενη ε, κυκλοφορίας σε δίκτυα ή σε κόμβους μεγάλης κίνησης, είτε πρόκειται για απαγορεύσει στην κυκλοφορία. Συμφωνώ, όπως και εσείς και χαίρομαι, που θεωρείται σημαντικό να δοθεί έμφαση στην ποιότητα περισσότερο και όχι στην ε, ποσότητα. Τα συστήματα ITS, τα εφή e, συστήματα μεταφορών είναι πολύ σημαντικά βεβαίως προκειμένου να ε, εξασφαλιστεί μια οικονομία οικολογικά αποτελεσματική. Και βεβαίως η νέα τεχνολογία πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα στις προτάσεις αυτές. Ο κύριος Λουίς Δεγκόντας Πασκουάλ έθεσε επίση μια ερώτηση για συνεργασία με άλλες χώρες. Δεν θέλει να υπογραμμίσω ότι η Σουηδική Προεδρία έχει συμμετάσχει στην ε, κατάρτιση του 18 ου προγράμματος μας με τη Γαλλική και τη Τσεχική Προεδρία, ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέχεια στο έργο αυτό. Συνέχεια απαραίτητη έτσι ώστε να ε, προχωρήσουμε αποτελεσματικά αλλά και να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία και με εσάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. πολλές από τις πρωτοβουλίες δε, που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. θα ε, δουν συνέχεια και από την Ισπανική Προεδρία με την οποία έχουμε επίσης την συνεργασία. Και πέραν της τελής συνεργασίας έχουμε τη φιλοδοξία να διατηρήσουμε ε, τον διάλογο Πρόεδρε, με συγχωρείτε που μακρύγορο τόσο. ο κύριος Άλβαρες, ρώτησε για ατυχήματα. Και βεβαίως λυπούμε για τα τραγικά αυτά ατυχήματα που έλαβαν χώρα. αεροπορικά ατυχήματα. Εξετάζουμε βέβαια ιδιαίτερα τους ε, λόγους για τους οποίους έγιναν τα ατυχήματα αυτά. Κοιτάμε τις μελέτες που θα εκπονήσουν οι ειδικοί. Και θα δώσουμε συνέχεια στην υπόθεση. Πρόεδρε, πιστεύω ότι έχω απαντήσει στις περισσότερες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Υπήρχε και ένα ζήτημα των αστικών μεταφορών η Επιτροπή έχει ε, προβλέψει ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, την οποία και περιμένουμε. Και με βάση αυτήν θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε για τις ε, μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι για την Σύμβαση των Άλπαιων. Βεβαίω, Πρόεδρε. Βεβαίω. Όπως είπα και νωρίτερα. συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο το σύνολο των εργασιών για την Σύμβαση των Άλπων και πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη που την έχουν υπογράψει συνεχίζουν ή που εμπλέκονται τέλο πάντων, συνεχίζουν το έργο τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τη συμβολή σας, τι συζητήσει μα σήμερα, τι παρατηρήσεις σα, αλλά και τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των ε, συναδέλφων. Πιστεύω ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα. Στη Στοκχόλμη έχουμε ένα ραντεβού σύντομα και σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Καλή επιτυχία στη Σουηδική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε λεπτά διάλειμμα συνάδελφοι και θα ξαναρχίσουμε μετά. Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Δεύτερη φορά σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να καθίσετε. Την τρίτη φορά που θα το πω δεν θα είναι εξίσου ευγενική η πρόσκλησή μου. Mr. Kolicek. Ξεκινώ. Όσοι θέλουν, όσοι θέλουν να έχουν παράλληλες συζητήσεις να το κάνουν απ' έξω. Ιδίως ε, στις ομαδούλες εκεί στα δεξιά μου. Κομισιόν, βουλευτές, υπάλληλοι. Το δύο φορές ήδη. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με, τον... με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορικών Μεταφορών, την ΕΑΣΑ, ιδίως δε τον Γενικό Διευθυντή, τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον κύριο Γκούντου, που κάθεται εδώ, δεξιά μου. Δεξιά σας. Εισαγωγικά, να πω τα εξή. Όπως ξέρετε θέλουμε να έχουμε τους επόμενους δύο μήνες συζητήσεις με όλους τους εκτελεστικούς διευθυντές των υπηρεσιών ασφάλειας. Ε, τον, τον παράλληλο μήνα θα δούμε τον υπεύθυνο για τις μεταφορές. Εσείς είστε ο κύριος υπεύθυνο της ασφάλειας στον αέρα. Όπως ξέρετε, πολλοί νέοι συνάδελφοι μπορεί να μην ξέρουν ούτε καν τι ακριβώς κάνει ο οργανισμός σας. Θα σας ζητούσε λοιπόν να μιλήσετε για ένα 15 λεπτό και μετά θα ακούσουμε σχόλια και ερωτήσεις των μελών. Σας ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για τη συμμετοχή σας ε, στην σημερινή συνεδρίαση. Έχετε το λόγο κύριε Κουντού. να έρθει στην πλατφόρμα ο κύριος στο βήμα ο κύριος Γκουντού. Θέλετε να έρθετε εδώ. Στο Προεδρείο κύριε Γκουντού, γιατί φαντάζομαι ότι η κυρία Φώστερ θέλει να βλέπει τι ομορφιές σας. Ένας λόγος που τον είχαμε εκεί τον κύριο Γκουντού ήταν ότι είχαμε εδώ τους ειδικοί δηλαδή πρόεδροι, οπότε τακτικά θεωρήσαμε είναι σκοπιμότερο να είναι μακριά τους. Τώρα που τον φέραμε πάνω ευχαριστημένοι όλοι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ που με καλέσατε στο βήμα αυτό. Τιμή μου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, όπως ήθιστε πάντα, είναι τιμή και χαρά για μένα να μιλώ στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και αναγνωρίζω κάποια οικία πρόσωπα από εδώ και από εκεί. Ξέρω ότι έχετε και νέα μέλη που δεν έχουν συμμετάσχει στον καρποφόρο πάντα διάλογο που είχαμε με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υποστήριξη που πάντα η Επιτροπή σας προσέφερε προς τον οργανισμό μου και για το ενδιαφέρον που δείχνει όπως και εμείς για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη. Θα επικεντρώσω την εισήγησή μου σε θέματα επικαιρότητα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο και για τα οποία παίζει και σημαντικό ρόλο. Πριν αυτό ωστόσο θα ήθελα εντάχει να σας αναφέρω τους πόρους σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και το προσωπικό που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τώρα. Γιατί βεβαίως το θέμα των πόρων είναι πάντα καθοριστικό. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, η υπηρεσία που όπως γνωρίζετε βρίσκεται στην κολονία, έχει 500 άτομα περίπου από όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη και μεταξύ αυτών η μεγάλη πλειοψηφία είναι έκτακτη υπάλληλη Μέχρι το 2010 θα απασχολεί περί τα 600 άτομα, άρα προβλέπουμε μια μικρή αύξηση ακόμα, μια κάποια αύξηση του προσωπικού. Ένα σημαντικό θέμα που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν δύο εκπρόσωποι μας ήδη στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ και την Κίνα, τη Washington και το Πεκίνο ειδικότερα. Νέοι εκπρόσωποι της, του οργανισμού θα προσληφθούν στο εγγύς μέλλον για να είναι παρόντες ε, στις μεγαλύτερες, στις πιο σημαντικές αερο πορικές περιοχές ε, ενδιαφέροντος αεροπορικού στον κόσμο. Προϋπολογισμός. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 2009 ήταν περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ. Θα αυξηθεί το 2010. Τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού αυτού προέρχονται από τα τέλη του βιομηχανικού κλάδου. Ένα τέταρτο από τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής στο θέμα αυτό και επαναλάβω αυτό που είπα στην προηγούμενη παρέμβασή μου στην Επιτροπή σας. Πιστεύω ότι σήμερα διαθέτουμε επαρκείς πόρους για να υλοποιήσουμε όθα τις αρμοδιότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, όπως ξέρετε, οι αρμοδιότητες αυτές θα επεκταθούν και θα επανέλθω αργότερα. Η υπηρεσία πρέπει να είναι σίγουρο ότι και μέσο και μακροπρόθεσμα θα διαθέτει, θα διαθέτει τους ε, πόρους για να λάβει τα νέα καθήκοντα που μπορεί να τις ανατεθούν. θα, αναφερθώ τώρα στην επέκταση των του οργανισμού που ψηφίσετε. Η πρώτη επέκταση των ευθυνών μας περιλαμβάνει νέα καθήκοντα στον τομέα της αεροπορικής εκμετάλλευσης, των αδειών πιλότων και των αδειών ε, ε, ε, οργανώσεων και επιχειρήσεων από τρίτες χώρες το χρονοδιάγραμμα τηρείται σε ό,τι αφορά αυτή την ε, επέκταση. Για, οι, δύο οι προϋποθέσεις για τις δύο πρώτες επεκτάσεις πλην αυτών των τρίτων χρόνο έχουν ολοκληρωθεί. Στη βάση που ο κανονισμό ε, στηρίζεται στον στην, στην υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα βασικά κάνοντα ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού τον αντίκτυπο που μπορούσε να έχει ένας νέος κανονισμός στις εμπλεκόμενες πλευρές. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των ορών πτήσεως. Όπως συμφωνήθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ζητήσαμε και δημοσιεύσαμε μια επιστημονική μελέτη για τον περιορισμό του χρόνου πτήσεως. Το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ε, δημιούργησαν ε, σοβαρές αντιρρήσεις από πλευράς και αεροπορικών εταιριών και συνδικάτων πιλότων. Οι αεροπορικές εταιρείε μάλιστα παραπολέθηκαν στον επίτροπο κ. Ταγιάννη. Εμεί αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής στις μελλοντικέ προτάσεις μας σε συνεργασία με την Επιτροπή και τις εμπλεκόμενες πλευρές. Παράλληλα, εξετάζουμε τη διαχείριση κινδύνου τη κόπωσης του πληρώματος που αυτή τη στιγμή αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερη προσοχή σε διεθνέ επίπεδο τόσο στο, στο, στο OACI και στον Διεθνή Οργανισμό Αεροπορικών Μεταφορών και στην Αμερικανική FAA. Θέλουμε να περιλάβουμε συστήματα διαχείρισης της κόμπωσης στα συνολικά συστήματα διαχείρισης ασφάλειας. γενική αεροπορία τώρα. Η υπηρεσία πάντα αναγνώρισε τη σημασία της γενικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Προσπαθεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξή της, ε, μειώνοντας τις διοικητικές, ε, τα διοικητικά βάρη του κλάδου, χωρίς να επηρεάσει την ασφάλεια. Η έννοια European Light Aircraft είναι παράδειγμα της πρωτοβουλίας αυτής. Το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή άδεια πιλότων αναψυχής προσπαθεί επίσης να αναζωογονήσει την γενική αεροπορία στην Ευρώπη. Βλέπετε λοιπόν ότι δραστηριοποιούμε στον τομέα αυτό. Δεύτερη επέκταση αρμοδιοτήτων τώρα, το τελικό κείμενο της οποίας θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η δεύτερη αυτή επέκταση στον τομέα της ασφάλειας και της εχείρησης των αεροπορικών μεταφορών, των υπηρεσιών αεροπορικής πλοήγησης και των αεροδρομίων. Η δουλειά προετοιμασίας έχει υλοποιηθεί. ιδίω συνεργαζόμαστε με το Eurocontrol για την μετάβαση, μετάπτωση μεταξύ των δύο συστημάτων. Το χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο. Συνολικά, για την πρώτη και τη δεύτερη επέκταση, η πόροι, η διάθεση των απαραίτητων πόρων είναι προπόθεση για, να, για την επιτυχή υλοποίηση των νέων καθηκόντων μας και στην πρώτη και στη δεύτερη επέκταση. Και βεβαίως χαίρομαι για την υποστήριξή σας όταν συζητηθούν λεπτομεριακά η χορήγηση, το θέμα των πόρων και η χορήγησή τους. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε κάποια θέματα επικαιρότητα στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορικής ναυσιπλοείας και θα ξεκινήσω με το πλαίσιο προστασίας των παιδιών. Είναι ένα θέμα που ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για κάποιους από εσάς, αλλά και για πολλούς γονείς παιδιών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Ο οργανισμός εξέτασε την κατάσταση προσεκτικά και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Δεν υπάρχει διεθνής πρακτική ενιαία σε ό,τι αφορά τη χρήση των ε, προστατευτικών ε, δομών για τα παιδιά. Ο κανονισμός EU Ops αφήνει στα εθνικά συστήματα την επιλογή των συστημάτων που εγκρίνουν. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούν μια, συμπληρωματική, μια επιπλέον ζώνη η οποία αφορά για την κοιλιά και το στομάχι για τη μεταφορά παιδιών κάτω από δύο έτη χωρίς να έχουν αναφέρει προβλήματα. Μία μελέτη που έγινε με βάση μετά από αίτημα του οργανισμού διαπίστωσε ότι στατιστικά υπάρχουν ευτυχώ λίγα στοιχεία που να δείχνουν ότι η πρακτική αυτή είναι επικίνδυνη. Η επιστημονική ανάλυση από την άλλη πλευρά αναφέρει ότι ε, υπάρχουν πλονεκ, πιθανά πλεονεκτήματα από τη δημιουργία θέσεων για παιδιά. Είναι σαφές ότι πρέπει να αναλάβει δράση ο οργανισμός και οι αεροπορικές εταιρείε πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν στα παιδιά να ταξιδεύουν με ειδικέ με ειδικά καθίσματα το ζητούν οι γονεί. Ωστόσο, καταρχά ο οργανισμό έχει πιστοποιήσει ένα ειδικό κάθισμα για παιδιά που χρησιμοποιείται από μία επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε από τον κλάδο να ε, επινοήσει νέα, ε, νέες, νέες κατασκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα. Δεύτερον, ε, ζητούμε από, τους, ε, από τις επιχειρήσεις να σκεφτούν τις συμπληρωματικές πληροφορίες όταν σχεδιάζουν τους νέους τύπους ε, καθισμάτων. Ζητήσαμε από όλους τους ευρωπαϊκούς, όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μας δώσουν τα σχετικά στοιχεία. Τρίτον, θα συζητήσουμε με τους διεθνείς εταίρους μας, ιδίως τον ΟΑΣΥ και την FAA για τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν τόσο ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιση προστασία των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως θα μπορούσαμε να προτείνουμε να υιοθετηθεί ανα πάσα στιγμή μια σειρά περιοριστικότερων μέτρων να διαπιστώσουμε ότι οι επιχειρηματίε ε, δεν θέλουν να συνεργαστούν. Τώρα, το ατύχημα της πτήσης Air France 447. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, πολλά αναφέρθηκαν για το τραγικό ατύχημα τη πτήση της πτήσης 447 τη Air France την 1η Ιουνίου φέτο. Μέχρι τώρα η έρευνα δεν εντόπισε την αιτία του ατυχήματος. Αυτό το επανέλαβε ξεκάθαρο ο διευθυντής ε, του Γραφείου Έρευνας και Ανάλυσης της Γαλλίας που ήταν υπεύθυνο για την ε, έρευνα αυτή. Ο οργανισμός συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε να βοηθήσει τους Γάλλους ερευνητές στους τομείς αρμοδιότητάς μας. Η συνεργασία μας με την ερευνητική ε, υπηρεσία είναι εξαιρετική. Επιπλέον, αναλάβαμε, λάβαμε και μια σειρά αποφάσεων και προληπτικών μέτρων. Στις 9 Ιουνίου ήδη, λίγε μέρε μετά το ατύχημα δηλαδή, ο οργανισμός δημοσίευσε ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ασφάλεια, ένα safety information bulletin δηλαδή, με επιχειρησιακέ συστάσεις. Μια λεπτομεριακή τεχνική ανάλυση αλλά και δοκιμές συνεχίζονται αυτή τη στιγμή σε σχέση με το, την, την, την ε, αντίσταση που δίνουν τα στοιχεία του αεροσκάφου σε μείωση ταχύτητας. ωστόσο, δεν θέλουμε να συνδέσουμε το ατύχημα με συγκεκριμένες ευθύνες χωρίς να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Θα ήταν πολύ ε, λάθος να κατηγορήσουμε οποιονδήποτε χωρίς να έχουμε στη θέση μας όλα τα στοιχεία. Ο ρόλος μας είναι να βελτιώσουμε την ασφάλεια τώρα και πάντα δεν υπαγορεύουμε τις αποφάσεις μας βάσει των στοιχείων των μέσων ή ομάδων πίεσης, αλλά σε αντικειμενικά κριτήρια. Η ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας σε κάθε δουλειά που κάνουμε, είτε μιλά για πιστοποίηση προϊόντων, είτε για νέους κανόνες που προτείνουμε. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι δεν κάνουμε νέες προτάσεις κανονιστικής ρύθμισης παρά μόνο είμαστε πεπισμένοι ότι ε, διαφυλάσσουν ή βελτιώνουν την ασφάλεια. Τώρα, Ποιο είναι το γενικό επίπεδο της, της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη. Ε, Α σταθούμε στα στοιχεία που έρχονται από τι δικέ μα αναλύσει που βασίζονται στην ε, ετήσια έκθεση για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών που σα καλώ να διαβάσετε. Από τα θετικά. Τα ατυχήματα που είχαν θανάτου στον κόσμο συνέχισαν να μειώνονται την τελευταία δεκαετία. Η Ευρώπη συνεχίζει να έχει ένα από τα καλύτερα επίπεδα ασφάλεια στον κόσμο. Αυτό ωστόσο δεν αρκεί. Είμαστε πίσω από τη Βόρεια Αμερική και με τα δύο ατυχήματα τη Πανέλ πέρσι και τη Φανς Φέτο, η τάση δεν είναι καλή. Θεωρώ ότι η διατήρηση ενό χαμηλού επίπεδου ατυχημάτων στις, ε, ε, στις εμπορικές μεταφορέ μεταφορές παραμένει ε, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μα. Για να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε στοιχεία. Κάθε ατύχημα πρέπει να αναφέρεται βάσει τη ευρωπαϊκή της Βλέπω ωστόσο δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, η, φυστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υλοποιείται παντού στην Ευρώπη. Δεύτερον, ο ρόλος του οργανισμού πρέπει να ενισχυθεί. Χρειάζεται να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα, ε, σκο, στοιχεία, <coughs> τα αναγκαία στοιχεία. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές πρέπει να οργανωθούν τόσο ώστε να αναλύουν από κοινού τα ατυχήματα. Η Επιτροπή προέβλεψε να ενισχύσει την σχετική νομοθεσία για την αναφορά ατυχημάτων και τα στοιχεία των δυστυχημάτων και σε αυτό το κείμενο θα διευκρινιστεί και ο ρόλος του οργανισμού, κάτι που είναι χρήσιμο και θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη. Επίσης, έχουμε όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των ανθρώπινων παραγόντων και του κρίσιμου ρόλου που παίζει ο άνθρωπος στην ασφάλεια. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να, δοθούν, να γίνουν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της ενημέρωσης του πληρώματος σκάφους. Η FAA συμφωνεί με την άποψη αυτή. Ο οργανισμός θα οργανώσει λοιπόν μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη για την κατάρτιση των πιλότων στις 24 Νοεμβρίου στην Κολομβία για να συζητήσει νέες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πέραν αυτού, σε συνεργασία με τον κλάδο, ο οργανισμός μας έχει ήδη δημιουργήσει ειδικέ ομάδες ε, εμπειρογνωμόνων για τις εμπορικές αερομεταφορές, το E-Cast για τη μεταφορά μέσω ελικοπτέρων, το οποίο αποκαλούμε E-Hast και την γενική αεροπορία, το EGAST, ούτως ώστε να υπάρξουν πρωτοβουλίε ασφάλειας σε κάθε έναν από αυτούς τους τρεις καθοριστικού τομεί: αεροπορικέ μεταφορές, ελικόπτερα και γενική αεροπορία. Πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίε αυτές αποτελούν μια πρώτη φάση για μια πιο σφαιρική στρατηγική. Δεν χρειάζεται να αντιδρούμε μόνο στον τομέα τη ασφάλεια αεροπορικών μεταφορών. Μετά από 6 χρόνια λειτουργία πρέπει να παίξουμε και έναν πιο ενεργό ρόλο. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική που θα βλέπει προ το μέλλον και συγκεκριμένου στόχου βελτίωση ασφάλεια. Είμαι πεπισμένο στην Ευρώπη έχουμε και τι γνώσει και του αναγκαίου πόρου για να γίνουμε μια ασφαλέστερη περιοχή στον κόσμο. Μετά με βάση τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού ε, Πολιτικής Αεροπορίας θα αναπτύξουμε μαζί με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ασφάλεια αεροπορικών μεταφορών. Το πρόγραμμα αυτό θα επιτρέψει να περιγράψουμε την οργάνωση τη ασφάλειας, ασφάλεια αεροπορικής στην Ένωση και τι δράσει που θα πρέπει να αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζοντα προφανώ ότι κάθε χώρα έχει και αυτή τι δικέ τη πρωτοβουλίε. Η ασφάλεια στην Ευρώπη, η ασφάλεια των ευρωπαϊκών μεταφορών στην Ευρώπη είναι ένα σύστημα στο οποίο θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι εταίροι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Εθνικέ κυβερνήσει, οι υπεύθυνε αρχέ και ο κλάδο. Ο οργανισμό θα προτείνει τη δημιουργία ενό πιλωτικού, μια ομάδα ε, καθοδήγηση του προγράμματο αυτού. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, το χρόνο που έχω στη διαθεσή μου προσπάθησα να υπογραμμίσω τι τωρινέ προτεραιότητε του οργανισμού. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα, πολλά άλλα πράγματα για άλλα ζητήματα. Ε, Ήδη από τώρα θέλω να εκφράσω τη χαρά για τι ανταλλαγέ και τι συζητήσει που θα είχαμε τα επόμενα πέντε χρόνια και ελπίζω να έχετε χρόνο να επισκεφτείτε τον οργανισμό μα στην κολονία όπου θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή σα και τα μέλη πιστεύω πως έχουν συμβολές να κάνουν εκ μέρους του Άλφ και ο Γκρός έχει το λόγο παρακαλώ ευχαριστώ για την παρουσία σας για την παρουσίασή σας και τις πληροφορίες που μας έδωσαν πιστεύω πως στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε ε, να συναντούμε θα στις Βρυξέλλες Νομίζω πως αυτό αποτελεί μέρος της δυνατότητας που έχει η δική μας Επιτροπή Μεταφορών να μπορέσουμε να επισκεφθούμε τις εταιρείε αυτές και το πρακτορία αυτά. Υπήρξε αυτή η πρώτη φορά μια πληροφόρηση και θα αρκεστώ σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά τον προϋπολογισμό. Αναφερθήκατε. Ξέρετε, το συζητήσαμε χθε και το ψηφίσαμε σήμερα το προπολογισμό και πέρα από τους αριθμούς που δώσατε εσείς προηγουμένως υποτίθεται από τους λίγους που λέτε αυτή τη στιγμή ότι είναι ικανά τα χρήματα τα οποία παίρνουμε υπάρχουν ε, τα λειτουργικά έξοδα, τα διοικητικά έξοδα πιστεύω είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό επίσης να αποφύγουμε σε ορισμένους ε, συναδέλφους τις προκαταλήψεις που έχουν και οι οποίες είναι υπερβολικές. Το δεύτερο έχει σχέση με την κατάρτιση. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα και είπατε ότι αντίθετα σε αυτά τα οποία ακούμε ή διαβάζουμε όσον αφορά το ατύχημα της Air France δεν οφείλεται στην κατάρτιση όσον αφορά τις δύσκολες συνθήκες είπατε αυτό το πράγμα αλλά στη συνέχεια είπατε ότι η εμπειρία σας ότι μπορεί να σας κάνει να κάνετε προτάσεις για την κατάρτιση. Αυτό έχει σχέση με τη βασική κατάρτιση ή τη συνεχή κατάρτιση. Και το τρίτο θέμα έχει σχέση με την ασφάλεια. Πιστεύω πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πάντα υποστηρίχθηκε σε αυτό το κοινοβούλιο και θέλω να ρωτήσω το εξή. Ποιο αντιτίθεται και τι αντιτίθεται όσον αφορά τη δυνατότητα να γίνει κάτι αυτή η ασφάλεια όλο και περισσότερο. Ή είναι οι πρωτοβουλίε ή τα προνόμια που έχουν τα κράτη-μέλη και οι διάφορε χώρε που έχουν και τα πρακτορία, οι εταιρείε ημένα αφενό και η δε αφετέρου. Κύριο Λάικφριτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Γκουντού, αυτό το οποίο παρουσιάσατε δείχνει ότι η εταιρεία σας είναι μια εταιρεία η οποία έχει πετύχει είναι επιτυχημένη και είναι κατά την άποψή μου αυτή που είναι πιο σημαντική καθότι ασχολείται με θέματα τα οποία είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικά που είναι, γι' αυτά είναι η ασφάλεια και επιτρέπει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αερίου χώρου. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα εσείς και βεβαίως είναι θέμα πώς μπορούν οι ικανότητες αυτές να επεκταθούν. Ε, δεν είναι αρκετές οι δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε με, δια της χρηματοδοτήσεως να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο, να γίνεται μια καλύτερη εργασία και πολύ πιο ποιοτική. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση και διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δηλαδή όλες οι, τα, τάσεις είναι οι αυτές ότι θα πρέπει οικονομία, οικονομία, οικονομία, εξοικονόμηση μάλλον θα να πούμε αυτό, υπενήσω αυτό. Και φρονώ πως αυτό είναι λαθασμένο διότι υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις οι οποίες θα γίνουν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πρέπει, θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το κίνδυνο που ελοχεύει ότι δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν οικονομίες σε αυτές τις εταιρείε οι οποίες αυτή τη στιγμή φτάνουν στο ΕΑΣΑ και εγώ θα ξανά ξέρω ποιες είναι οι ιδέες τις οποίες εσείς μπορείτε να πτήσετε όσον αφορά αυτή την αντίσταση όσον αφορά την εξοικονόμηση. Επίσης θα ήθελα να ξέρουμε για το ατύχημα της Πανέρ που έχει γίνει είχαμε την εντύπωση βλέποντας αυτά τα, τα εξωτερικά βλέπουμε ότι οι Ισπανικές αρχές με την Άιζα δεν είχαν πάρα πολύ καλή επαφή και πάρα πολύ συνοντισμό και είχε μία έλλειψη ενημέρωσης και εν τελική αναλήψη τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα έπρεπε να εξελίχθουν. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν κατά πόσον υπήρξε πρόβλημα από τη δική σας σκοπιά όσον αφορά την ασφάλεια και τι μπορεί να γίνει καλύτερο στο μέλλον από το θέμα του αυτού. Σε σχέση με αυτό ακόμη στο θέμα των ατυχημάτων επιμένω και λέω κατά πόσο στα πλαίσια της ευρωπαϊκών, των ευρωπαϊκών εταιριών ποιες είναι εκείνες οι οποίες είναι λιγότερο ασφαλείς. Το τρίτον, κατά πόσον ο νομοθέτης έχει αποφασίσει κατά πόσον ο θάλαμος του αεροπλάνου θα είναι κοινό και πώς ακριβώς οι διάφορες εταιρείες αντιδρούν σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η, από τους φιλελεύθερους η κυρία παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Γκουντού για την παρουσίαση της. Υπάρχουν εδώ νέα πρόσωπα τα οποία δεν τα γνωρίζετε. Εγώ είμαι μόλις εξελέγει και έχω ερωτήσει πάρα πολύ σαφείς και σχέση με την κατάρτιση. Είπατε προηγουμένως όσον αφορά την ασφάλεια. Χρειάζονται βελτιώσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Πιστεύω πως νομίζω στα πλαίσια της κατάρτισης η ασφάλεια είναι εκ των για τα αεροπλάνα και πολύ συγκεκριμένοι οι Αμερικάνοι είναι καλύτερα. Αλλά ποια είναι αυτά τα οποία λείπουν, ποια είναι η λήψη οι οποίες έχουμε εμείς σαν Ευρωπαίοι, ούτω ώστε η ευρωπαϊκή ε, μεταφορά να γίνει πολύ καλύτερη. Ο εκπρόσωπο των Πρασίνων παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Όσον αφορά τις, τα καθήκοντα των παιδιών, είναι κάτι το οποίο παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και ευελπιστώ πως μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, σε μια, να καταλήξουμε στην υπόθεση όσον αφορά την καλύτερη ασφαλειά τους. Είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν πολύ, πολλές λίγες περιπτώσεις, αλλά ωστόσο θα πρέπει να δούμε ότι σε διεθνές επίπεδο, στις στατιστικές οι οποίες έχουμε, βλέπουμε αυτοί οι οποίοι δεν φορούσαν κατά τη διάρκεια του ζώνες τους και δυστυχώς δεν φαίνονται ορισμένες φορές όλα αυτά τα στοιχεία στην στατιστικές που έχουμε αναχείρας. Ξέρω ότι η δικασία είναι περίπλοκη και για όλους και υπάρχουν λίγες προτάσεις οι οποίες γίνονται. Αυτό είναι πολύ σαφές στο μυαλό μου. Ωστόσο πιστεύω εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ούτω ώστε να προχωρήσουμε με πολύ λιγότερες δυσκολίες και να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε τους γονείς πιστεύω εντάχει να πούμε πολύ, ε, πολύ σωστά ότι αυτή η κυλιακή και στομαχική αν θέλετε ζώνη μπορεί να είναι λυτρωτική σωτήρια σε ορισμένε περιπτώσεις και οι μελέτες οποίες έχουμε αναχείρας έχουν μερικές επιλογές. Θα πρέπει όμως στο, μένος, στο μέλλον να υπάρχει ένα προσαρμοσμένο κάθισμα για τα παιδιά, για τα πολύ παιδιά και σε περίπτωση πτώσης ή ατυχήματος όταν υπάρχει ατύχημα δεν μπορεί η μητέρα να πάρει το παιδί στην αγκαλιά τη. Δεν επιτρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και διαρωτώ με κατά πόσο εσεί μπορείτε να γνωρίσετε, να αν υπάρχει δυνατότητα μιας πολύ ταχείας διαδικασίας ούτως ώστε να γίνει κάτι τέτοιο και είμαι απόλυτα πεπισμένη πως αυτό μπορεί να επεκταθεί από την Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα το οποίο ήταν σε διεθνές επίπεδο και σε αυτό το σημείο η διεθνή ευαισθησία είναι παρούσα και όλοι ζητούν να φτάσουμε σε ένα απτό αποτέλεσμα. Δύο ακόμη μικρά πραγματάκια που δεν είναι καθόλου μικρά βεβαίως στο οργανόγραμμα βλέπω γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία άπτονται του το θεμάτων του περιβάλλοντος. Κατά, τι, με τι ασχολούνται, ποιε είναι η, η απασχόλησή τους. Και κάτι ακόμη το δεύτερο, την γεμενική εταιρεία, αεροπορική εταιρεία. Ξέρετε ότι η ΑΕΡ έχει το δικαίωμα να προσγειωθεί στη Γαλλία. Τι συμβαίνει με τι άλλε χώρε, υπάρχει κάποια αντίστοιχη απαγόρευση. Βλέπουμε δυσκολίε και ποιε είναι οι προοπτικέ όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετώ τον κύριο Κουντού και χαίρομαι που είστε εδώ. Έχουμε συζητήσει. Είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα από την 2009 και 2004 και πιστεύω πως η εταιρεία το έχει κάνει πάρα πολύ ε, καλή εργασία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία τίθενται και θα θέλουν να τα θέσω. Δεν νομίζω πως πραγματικά μας διέφυγαν αυτά τα θέματα. Το πρώτο είναι όχι μόνο για σας, αλλά για την Επιτροπή εδώ παρούσα. Και έχουμε τεράστιες ευθύνες όσον αφορά πραγματικά πώς εσείς χρηματοδοτείτε, δομικά Ωστόσο, είπατε ότι τα τρία τέταρτα του προπολογισμού έρχονται από συμβολές και από τέλη τα οποία υπάρχουν και το ένα τέταρτο έρχονται από εμά. Υπάρχει ένα σαφές θέμα ότι μακροχρόνια η χρηματοδότηση θα πρέπει να δούμε χρόνο με χρόνο πραγματικά τι γίνεται και υπάρχει μια αύξηση αλλά δεν πραγματικά πώς θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο εδώ σε αυτό το θέμα της αυξήσεως διότι παίρνονται για τα ATM την, τον, έλεγχο, τον έλεγχο των αεροπορικών το, και άλλα θέματα. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες και αυτά όμως που κάνετε αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερα αυξάνεται η αρμοδιότητά σας και θα πρέπει να ξέρουμε πώς χρηματοδοτήσετε, θα πρέπει να έχουμε ένα δεκαετές πρόγραμμα για να ξέρουμε ποιος πληρώνει, πώς πληρώνει και γιατί. Ανησυχούμε λοιπόν πραγματικά το μεγαλύτερο ποσοστό έρχεται από την βιομηχανία. Αλλά αυτό εάν δεν πηγαίνει καλά, τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τα εισοδήματα τα οποία παίρνουν έρχονται από εκεί. Είναι ένα θέμα να το σχολιάσετε, γιατί εγώ να το σχολιάσετε αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα ήταν το θέμα το οποίο τέθη όσον αφορά το περιβάλλον. Βεβαίω είστε ένας οργανισμός ασφαλείας. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι υπάρχουν επιπτώσεις από το περιβάλλοντος και το τελευταίο εάν πραγματικά βλέπετε το θόρυβο της εκπομπές κλπ εάν δείτε το NPA βλέπετε οι οποίες είναι αποφάσεις οι οποίες ακαλύπτουν τους πάντες και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ο ρόλος αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι μόνο η ασφάλεια και είναι και αυτό το θέμα και ακόμη δύο ερωτήσεις πρόεδρε αν μου επιτρέπετε επόμενο σημείο για τις σχολές, σχολές ε, εκμάθησης ε, πιλοταρίσματος. Αυτό το θέμα το, πρέπει να δούμε αυτό το θέμα, διότι είναι, υπάρχει ανησυχία για αυτό το θέμα. Και βεβαίως τα ατυχήματα που δημιουργούνται από αυτές τις μικρές σχολές και με αυτά τα μικρά αεροπλάνα, κατά πόσον πραγματικά έρχεται είστε ανεξάρτητος οργανωτικός, δεν πολιτικά, δεν υπάρχει πολιτική εμπλοκή και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τα τυχήματα τα αεροπορικά να αποκτήσουν μια πολιτικό, πολιτική χρειά. Θα ήθελα λοιπόν να μας διαβεβαιώσετε πως πραγματικά ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτική πτυχή η οποία εμπλέκεται διότι υπάρχει τα επόμενα ε, τα προηγούμενα έξι χρόνια υπήρχε ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο ιδιαίτερα ετέθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριο Σκόλιτσεκ από την Ενωμένη Αριστερά παρακαλώ και λίγα λεπτά για τους άλλους παρακαλώ. Πολύ σύντομα θα το εκτιμήσει ιδιαίτερη ιδιαίτερη Προεδρία. Πάντα ήμουν ακριβής και πάντα πολύ σύντομος όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία θέτω. Καλημέρα σας κύριε Γκούντου. Αν... Έξι Εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα τελευταία ατυχήματα έδειξαν ότι κάποιοι πιλότοι δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν το αεροσκάφος όταν σταματούν οι κινητήρες. Έχετε κάποιο πλάνο, κάποιο πρόγραμμα να βοηθήσετε την κατάρτιση των πιλότων για τέτοιες περιπτώσεις. Δύο. Η τυποποίηση των ελαφρών, των ελαφρού τύπου αεροσκαφών. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να υπάρξει μια τέτοια τυποποίηση στην Ευρώπη. Υπάρχει δυνατότητα και ανάποψη συντονισμού των δοκιμών ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σκάφη βάρους κάτω των 600 κιλών. θα μπορούσαν αυτά τα τεστ να μην γίνονται μόνο στην ΕΑΣ αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν εθνικές αρχές στις χώρες που κατασκευάζουν τέτοια έδρος σκάφη και τα περισσότερα είναι ευρωπαϊκά, έχουν τη δυνατότητα Επίσης, άτομα με αναπηρίες στις αερομεταφορές. Θέλετε, προτίθεστε να θέσετε κάποια πρότυπα για τα νέα αεροσκάφη ώστε να είναι προσπελάσιμα ε, για άτομα με αναπηρίες διότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, ένας ανάπηρος με καροτσάκι δεν μπορεί πρακτικά να μπει στο αεροπλάνο. Είπατε ότι θέλετε να έχετε 600 άτομα προσωπικό. Ο πίνακας που έχουμε μπροστά μας δίνει αύξηση 54 ατόμων στην Επιτροπή Προπολογισμών. Και εμεί σα δώσαμε τον προπολογισμό που μα ζητήσατε. Αρχικά, ωστόσο, μιλούσαμε για 447, όχι 600 μέλη προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τα υγρά και τα ζέλ στο, στα Θα κάνετε κάτι, κάτι γι' αυτό. Ο κύριος Χεσεμπόφσκι είχε συζητήσει μαζί μας και έλεγε ότι είναι ηλίθιο, άσχετο να υπάρχουν τέτοια όρια. Έχετε κάποια προγράμματα, κάποιες ιδέες σχετικά. Επίσης, θα υπάρξει κάποια περικοπή για τις μικρές εταιρείες όταν φτάνουμε στις δοκιμές. Κύριε Κουντού, μπορείτε να απαντήσετε σε κανένα λεπτό αν γίνεται. Γιατί έχω πολλούς άλλους που θέλουν να μιλήσουν. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις πάντα στον οργανισμό, αλλά τώρα 7 λεπτά για τόσες απαντήσεις δύσκολο. Να ξεκινήσω από την ερώτηση του κύριου Γκρός για τον προπολογισμό. Προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε και όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι αντίστοιχοι οργανισμοί με την Επιτροπή Προπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Εδώ και χρόνια και δύσκολα το καταλαβαίνω. Οι διαφορές μεταξύ λειτουργικών και επιχειρησιακών δαπανών. Ο κοινοτικό προπολογισμό έχει πέντε μεγάλους τίτλους, τρεις σημαντικούς δηλαδή, λειτουργικούς και ε, προσωπικό και συχνά οι οργανισμοί κατηγορούνται ότι έχουν, ότι έχουν δαπάνες λειτουργίας μικρές σε σχέση με το γενικό προπολογισμό. Πρέπει να σας πω ότι όταν έχω προσωπικό που δουλεύει ως διοικητικ... για διοικητικά καθήκοντα, το προσωπικό αυτό πληρώνεται από τον τίτλο 1. Αυτό που χαρακτηρίζεται εσείς ως διοικητικό κόστος, αλλά είναι επιχειρησιακές δαπάνες στην πράξη. Αν θέλετε να αυξήσω τις επιχειρησιακές σε σχέση, τις λειτουργικές σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες, θα πρέπει να κάνω outsourcing όλες αυτές τις δραστηριότητε, το οποίο είναι παράλογο. Θέλω λοιπόν να προσπαθήσω να εξηγήσω ότι η δομή σε τρεις τίτλους δεν είναι ουσιαστική για να καταλάβουμε αν οι δαπάνες, οι σχετικές δαπάνες είναι λειτουργικές ή διοικητικέ στους οργανισμούς. Ο, ο πρώτος και ο δεύτερος τίτλος είναι αυτός που περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες των οργανισμών. Πολλά ερωτήματα τέθηκαν σε ό,τι αφορά την κατάρτιση οι πιλότοι έχουν ένα πολύ περίπλοκο και σύνθετο ρόλο, ιδιαίτερα στην, στις εμπορικές μεταφορές που αντιμετωπίζουν τώρα όλο και πιο αυτοπανετοποιημένα αεροσκάφη. Τους ζητούμε να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις σχετικά σπάνιες. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι ένας πιλότος ο οποίος έχει μόνιμη βοήθεια αυτόματων μηχανημάτων πρέπει να είναι ικανός όταν τα μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν να πιλωτάρει ο ίδιος. Δεν θέλω να προδικάσω τα αποτελέσματα των, της διάσκεψης που θα έχουμε στις 24 Νοεμβρίου. Φαντάζομαι ωστόσο ότι η συνεδρίαση αυτή, το συνέδριο αυτό θα οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι κάποιοι θα κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αρχική κατάρτιση των πιλότων, η βασική κατάρτιση δηλαδή, και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να επέμβουμε στην κατάρτιση, ώστε η διαχείριση των εξαιρετικών περιπτώσεων, γιατί περί αυτών πρόκειται, να είναι πάντα στο μυαλό των πιλότων. Αυτό είναι πάντα κάτι, είναι κάτι που θεωρούμε ουσιαστικό. Ατυχήματα και συνεργασία με τα, τις ερευνητικές υπηρεσίες για τα ατυχήματα. Υπογράμμισα ότι η συνεργασία με τη γαλλική ε, με τη Γαλλική Αρμόδια Επιτροπή στην πτήση 447 της ΕΦΑΣ ήταν εξαιρετική. Αυτό δεν, ήταν, δεν συνέβη για το ατύχημα της Πανέρ. Χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να βρούμε τις σχέσεις. Προφανώς ο οργανισμός μας δεν είναι μια οργάνωση που ερευνά ατυχήματα. Εγώ θέλω να, είναι, να υπάρχουν ανεξάρτητοι ερευνητέ, αλλά ω πιστο, οργανισμός πιστοποίησης των αεροσκαφών μπορούμε να προσφέρουμε στους ερευνητέ τις γνώσεις που ε, προέκυψαν στη ζωή άλλων αεροσκαφών και άρα προσθέτουμε νομίζω μια ξεκάθαρη προστιθέμενη αξία. Από την άλλη πλευρά Όταν γνωρίζουμε καλά τι βρέθηκαν από την πραγματογνωμοσύνη, την έρευνα, μπορούμε να αναλάβουμε μέτρα, μερικέ φορέ επίγοντα μέτρα, για να βελτιώσουμε ή να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών. Και γι' αυτό λέγω απερίφραστα ότι δεν θέλουμε εμεί να είμαστε επιθεωρητέ ή ερευνητέ του οποιοδήποτε ατυχήματο. Δεν είναι η δουλειά μα αυτή, ούτε και πρόκειται να γίνει. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία των πραγματογνώμων, πραγματογνωμόνων. Θέλουμε όμω να έχουμε και αρκετέ πληροφορίε και ενημέρωση ώστε να κάνουμε τη δουλειά τη δική μα που είναι η βελτίωση του ενεργού μεταφορών. Έχουμε ένα business plan τώρα για τη χρηματοδότηση, πενταετές. Επιχειρησιακό πρόγραμμα, σχέδιο. Οι εισφορές θα εξασφαλίσουν ισοσκέληση του προϋπολογισμού μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορέσουμε διαπραγματευόμενοι με εκείνους με τους οποίους θα ζητούν τις υπηρεσίες μας, να προσδιορίσουμε το τιμολόγιο που ζητούμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά που αναλαμβάνουμε. Σε περίπτωση κρίσης τώρα τι κάνουμε. Τώρα διερχόμεθα μια πολύ σημαντική και για την αεροπλοεία κρίση Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα, έχουν μειωθεί σημαντικά τα ποσοστά πληρότητας των αεροπλάνων. Υποφέρουν από έλλειψη πληρότητας οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν πάνε καλά οι αεροπορικές εταιρείες, το γνωρίζουμε αυτό. Τούτου τουλάχιστον όμως την, την κρίση αυτή την διέρχεται τώρα ο αεροπορικός κλάδος χωρίς πρόβλημα ως προς τα πιστοποιητικά ε, ασφάλειες. Δηλαδή εξακολουθούν να μας ζητούν οι κατασκευαστές πιστοποίηση του υλικού τους που άλλωστε είναι και ο κύριος πόρος εσόδων για την υπηρεσία μας. Βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τις μικρές επιχειρήσεις των οποίων ορισμένε κλείνουν. Εάν μπορέσουμε λοιπόν σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να βρούμε ένα πολύ πιο μόνιμο, σταθερό τρόπο ε, χρηματοδότηση για την υπηρεσία μας, θα είμαι ευτυχής. Σε θέματα περιβάλλοντος τι κάνει η υπηρεσία μας, όπως το υπογράμμισε και η κυρία Λεχτεμπέργκερ. Έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται ειδικά με τις πτυχές της περιβαλλοντικές στην υπηρεσία μας. Με καθήκοντα πρώτον ρυθμιστικά, έχουμε δραστηριότητα σε επίπεδο Επιτροπής ΟΑΣΕ που ονομάζεται ε, CAO που ονομάζεται ΚΑΕΠ και σε επίπεδο Montreal ΟΑΣΕ έχουμε την προσαρμογή στην νομοθεσία, στις διατάξεις αυτές. Γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον. Στηριζόμαστε στην ICAO. Επίσης για το περιβάλλον, πιστοποίηση των προϊόντων. Που ξέρετε ότι έχουμε αναλάβει την πιστοποίηση των αεροσκαφών όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων και θορύβου. Οι δύο δραστηριότητές μας είναι αυτές που σας ανέφερα λοιπόν ως προς την, στο περιβάλλον και βέβαια η ΚΑΟ έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Υγρά και γέλες. Είναι ζήτημα ασφάλειας. Είναι ζήτημα ασφάλειας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε και είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή έχει αναλάβει να επιλύσει. Αφήνουμε αυτή τη δουλειά στην Επιτροπή. Δεν ασχολούμεθα εμείς με τα υγρά και τι γέλε που άλλωστε ξέρετε ότι και εμά όταν είμαστε επιβάτε, όταν έχουμε τον ρόλο του επιβάτη, πάλι μα δημιουργεί δυσκολίε. Ο Πρόεδρος. Επτά συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα παρακαλώ, για να δοθεί και απάντηση στις ερωτήσεις σας. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κύριε Διευθυντά για να σας ευχαριστήσω για τα πολύ ενδιαφέροντα σας λόγια και για την πολύ καλή διάθεση που δείχνατε πάντοτε απέναντι, της, απέναντι στην Επιτροπή μας. Όντως, λίγες είναι οι υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες διευρύνθηκαν τόσο πολύ και τόσο γρήγορα όσο αυτές τις δικής σας και σας ε, πείθει πιστεύω αυτό το γεγονός για το πόσο σημαντική θεωρεί την ασφάλεια των αερομεταφορών μεταφορών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα τελευταία τραγικά δυστυχήματα βλέπουμε πόσο απαραίτητο είναι η Ευρώπη να συνεχίσει να εργάζεται στον τομέα αυτό και στις ε, αερομεταφορές με τη χρυσή συζήτηση για τον προπολογισμό και όπω είπε και πολύ καλά η κυρία Φώστερ νωρίτερα, το αναφέρατε άλλωστε και εσεί, βλέπουμε ότι πρέπει οι πόροι που έχει στη διαθεσή τη η ΕΣΑ να είναι λυσμένοι να, να ε, ανέρχονται στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων που τις έχουμε αποδώσει. Το είπατε και εσείς και εμείς επίσης από την Επιτροπή των Μεταφορών θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε για το στόχο αυτό έτσι ώστε η υπηρεσία σας να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της σε αγαστές συνθήκες και να προστατεύει έτσι την ασφάλεια ε, των συμπολιτών μας. Η κυρία Άλβαρες. Όσο δεν πείσετε, μας σας παρακαλώ. Μα βέβαια, μα βέβαια. Πρώτον, να εκφράσω ό,τι καλύτερο στον κύριο Κουμπουντού για τη δουλειά του και τη δουλειά του οργανισμού του. Και να πω ότι πιστεύω πως πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του οργανισμού και ο διπλός συντονισμός με, όλη με όλο τον κλάδο της αεροναυπηγικής βιομηχανίας και των αεροπορικών μεταφορών. Ξέρω τις δυσκολίες που υπάρχουν στον τομέα αυτό και θα ήθελα να ακούσω την άποψή για τις συστάσεις που έκανε η Ισπανική Επιτροπή ε, ατυχήματο σε σχέση με το ατύχημα στην Ισπανία που τη Σπανέρ 6-7 προτάσεις έκανε, πέντε από τις οποίες αναφέρονται και στον οργανισμό, ενώ οι άλλες αφορούν άλλους οργανισμούς. Ο κ. Βαντέλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κανονισμός της υπηρεσίας σας προβλέπει και χρόνο ανάπαυσης, χρόνο εργασίας με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όταν όμως βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται διαρκώς ο χρόνος εργασίας ε, ή αν θέλετε είναι πιο αυστηρές διατάξεις περί χρόνου ανάπαυσης. Του αντίον βλέπουμε ότι στις εναέρειες μεταφορές ε, διαρκώς παρατείνεται ο χρόνος εργασίας των πληρωμάτων. Βλέπετε η αν θελετε ειναι πιο αυστηρες διαταξεις περι χρονου αναπαυσης τουναντιον βλεπουμε οτι στις αυτή να είναι ικανοποιητική. Μέσα σε ένα χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη κακή για μας. Ένα άλλο ζήτημα, η ασφάλεια των εναέριων μεταφορών είναι υψηλή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δύο μελανά σημεία θα σημειώσω. την ε, άφηξη ε, αεροσκαφών είτε από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες είτε από τις χώρες Αφρικής και τα υπερελαφρά αεροσκάφη. Ερωτώ λοιπόν για τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή για τις χώρες της Αφρικής έχετε, το... έχετε πρόθεση να επιβάλλετε διατάξεις και ε, συνθήκες αντίστοιχες με αυτές που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες διότι είναι βέβαια σοβαρό πρόβλημα η ασφάλεια που κινδυνεύει από τα αεροσκάφη αυτά. Ο κύριος Δηγράντες Πασκουάλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις. Ίσως κάτι να μην κατάλαβα καλά. Βέβαια. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξή: Ποια είναι η σχέση, οι διαφορές αν θέλετε μεταξύ του δυστυχήματος της Air France και της Pan Air. Ποια είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση των δυστυχημάτων αυτών μεταξύ των δύο ε, εθνικών αρχών και ούτω καθεξής. Ένα άλλο ζήτημα, ε, βέβαια δεν ξέρετε ότι όλους μας απασχολεί πάρα πολύ, το ζήτημα της κατάρτισης των πληρωμάτων, πιλότων κτλ. Συχνά ύστερα από ένα ατύχημα διαπιστώνεται ότι ε, οφείλεται το ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο αυτό λάθος, το οποίο μπορεί να έχει τεράστιες και τραγικές συνέπειες. Φυσικά μπορεί κάποια προβλήματα να πηγάζουν και από διοικητικά σφάλματα, αλλά συχνά διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανθρώπινο σφάλμα. Ερωτώ λοιπόν, εσείς βλέπετε ελλείψεις ως προς την κατάρτιση των κυβερνητών ή ε, μια επιπλέον ερώτηση, θεωρείτε ότι η επέκταση των εταιριών χαμηλού κόστους επιδεινώνει το επίπεδο, ρίχνει το επίπεδο της κατάρτισης των κυβερνητών στα αεροσκάφη που πετούν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιάλα Σάντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Φιτά για την παρουσία σας και να σας συγχαρώ για την, για εισήγηση που μας παρουσιάσατε. θέλω Κάποιες διευκρινήσεις και για την ε, Air France όμως να γίνουν. Βλέπετε εδώ ότι είμαστε πολλοί Ισπανοί ε, ευρωβουλευτές και προφανώς μας ενδιαφέρει περισσότερο το ε, δυστύχημα της Spanner. Θα ήθελα να ξέρω πώς μπορεί ο οργανισμός σας να βοηθήσει να προσφέρει μια ευρωπαϊκή διάσταση και να μας σχολιάσει τι έγινε μετά από την, το ατύχημα αυτό. Μιλήσατε για την εμπειρία της Ισπανίας που είναι σημαντική και για να μπορέσουμε να δούμε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος αυτού μια σειρά διαστάσεων που θεωρήσαμε σημαντικές το ότι οι αρχές ε, να διαθέτουν αμέσως τον κατάλογο των επιβατών που γενικά δεν ε, δίνουν, αλλάζουν οι εταιρείε τελευταία στιγμή, ξέρετε φεύγει κάποιο, δεν έχετε κάποιο άλλο. Επίση, είπατε ότι βρισκόμαστε μια μεταβατική φάση μεταξύ Eurocontrol και ASA και ότι έχετε ένα φιλόδοξο σχέδιο. Θέλω να ξέρω λίγο περισσότερο τι, τις Επίση, Επίσης μπορείτε να μα πείτε κάποιε λεπτομέρειε για τον τρόπο με τον οποίο η ASA θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κόπωσης του πληρώματος που θεωρούμε καθοριστικό αυτή τη φάση της επέκτασης των αεροπορικών μεταφορών. Κ. Μαρινέσκου. Μία ερώτηση. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με την ΆΣΑ και με τις νέες ευθύνες που θα έχει όταν αλλάξει ο κανονισμός. Επίση, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Μέσω της δουλειά σα ε, δίνετε πιστοποίηση σε αεροσκάφη, σε εξοπλισμό, σε προσωπικό, σε αεροδρόμια. Κάποια προβλήματα στη διαδικασία πιστοποίησης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να μετέχετε στην έρευνα ατυχημάτων γιατί εμπλέκεστε στην πιστοποίηση των αεροσκαφών. Και μία ερώτηση για το EU Ops. Όπως ξέρετε, πήρε 40 χρόνια να λειτουργήσει. Λόγω του ότι οι κοινωνικοί εταιρείε μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τώρα, μετά από 40 χρόνια, βρέθηκε σε μία θέση. Ε, έχει αρχίσει να λειτουργεί λιγότερο από 12 μήνες και τώρα φαίνεται ότι προσπαθούν να, να, να αλλάξουν τη λειτουργία του. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι μήπως θα ήταν σκόπιμο να υποστηρίξουμε το σχέδιο αυτό, να του δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο λειτουργία και μετά να προχωρήσουμε στην ανάλυση του κειμένου. Δεν θα συμφωνώ ότι ήταν να αλλάξει κάτι στην, ε, στο συγκεκριμένο υποτμήμα του Υγειού οπς θα έπρεπε να εμπλακεί και το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής όπως και η πρωτογενής νομοθεσία. Έχετε το λόγο. Άλλη μια μεγάλη πρόκληση να απαντήσω. Καταρχάς ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όλους τους βουλευτές που εξέφεραν την υποστήριξη στο πρόσωπό μου και το ρόλο της υπηρεσίας και την εκτίμηση για την παρουσία μας εδώ. Θα επαναλάβω ότι αν με προσκαλείτε πιο συχνά θα έρχομαι και πιο συχνά γιατί θεωρώ απαραίτητο να διατηρούμε το διάλογο αυτό. Δύο ουσιώδους χαρακτήρα τύπους ερωτήσεων άκουσα πρώτα απ' όλα τα ατυχήματα, σπάνια αφενός Air France αφετέρου, πώς αντιδρούμε σε κάθε, στην κάθε περίπτωση ή τι είδους αντιδράσεις εκδηλώθηκαν. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις σχέσεις της υπηρεσίας του οργανισμού ε, αφενός και όχι τις αρχές, τις εθνικές αρχές αφετέρου, αλλά τους ε, πραγματογνώμονες που ευερτίζονται με τη διερεύνηση του ατυχήματος. Προσπαθούμε λοιπόν να πτήσουμε επικοδομητικό διάλογο με τους πραγματογνώμονες αυτούς. Δύσκολο ήταν, πρέπει να σας πω στην αρχή, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά η περίπτωση της Πάνερ ήταν ακόμη σε οριακό, θα έλεγα, επίπεδο. Δηλαδή τον Αύγουστο του 2008 Ήμασταν διατεθειμένοι εμείς, ε, θα έλεγα, την ίδια ημέρα ακόμη να αναπτύξουμε την επικοινωνία και τις επαφές με, ε, ε, με την Ισπανική Υπηρεσία. Είχα ήδη δύο έτοιμους συναδέλφους να πάνε στην Ισπανία και να συνεργαστούν με τις Ισπανικές Αρχές, αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Καθυστέρησαν οι προσκλήσεις και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μας των σχέσεων τη υπηρεσία μας με τις αρχές διερεύνηση των ατυχημάτων. Τουναντίον, στην περίπτωση του ατυχήματο τη Air France και με τι επαφέ που είχαμε με την αντίστοιχη υπηρεσία διερεύνηση του ατυχήματο, είχαμε άμεση εμπλοκή ε, και χωρί καθυστέρηση μπορέσαμε να συμμετάσχουμε στη διερεύνηση του ατυχήματο. Πολύ διαφορετικό τρόπο δηλαδή ε, συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται νέο νομοθέτημα για τα αεροπορικά δυστυχήματα που θα διευκρινίζει και ποιο ρόλο θα έχει να διαδραματίσει η υπηρεσία μας γιατί μέχρι τώρα νομοθεσία βέβαια ε, δεν είχε προβλέψει την μεταγενέστερη άλλωστε ίδρυση της, ε, του οργανισμού μας. Για τον κύριο Μαρινέσκου θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν έχουμε ρόλο και εμπλεκόμενου μέρους και κριτή της υπόθεσης. Εμείς τις πληροφορίες θέλουμε να έχουμε με βάση ε, τα στοιχεία που έχει και το ε, πρότυπο του πιστοποιητικού και να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε μέτρα το ταχύτερο δυνατό. Γιατί αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό ε, να αναλαμβάνουμε δράση. Όχι, δεν κρίνουμε εμείς, δεν εμπλεκόμαστε εμείς κατά αυτό τον μεροληπτικό τρόπο. Πρέπει να, αφήνουμε ε, να κάνουν τη δουλειά τους οι ε, πραγματογνώμονες που επιλαμβάνονται της έρευνας. Κατάρτιση. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τη λειτουργία των υπηρεσιών χαμηλού κόστους ε, δεν αποδεικνύουν ότι έχουν χειρότερο επίπεδο ασφάλειας, του αντίον θα έλεγα σχεδόν, έχουν πολύ καλό επίπεδο ασφάλειας και οι εταιρείε low cost. Οι διαφορέ είναι διαφορετικού χαρακτήρα περισσότερο περισσότερο. Έχουν να κάνουν ε, τα προβλήματα στα, με τα νέα αεροπλάνα, τους αυτοματισμούς που είναι ενσωματωμένοι στο αεροπλάνο και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσει ο κυβερνήτης την ώρα που δεν θα ανταποκρίνεται ο αυτοματοποιημένος αυτός μηχανισμός στις εντολές του. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιλύσουν οι, ε, αεροπορικές εταιρείε μαζί και με τους κατασκευαστές των αεροπλάνων ε, για να βρεθεί η λύση. Και επίσης, εν τέλει, ως προς το χρόνο εργασίας, Έχει επιτευχθεί σε επίπεδο Κοινοβουλίου και Συμβουλίου συμφωνία ως προς το τμήμα Q με συνοδεία μιας επιστημονικής μελέτης, μιας πραγματογνωμοσύνης που θα, πρέπει να που θα έπρεπε να έχει αναθέσει η Επιτροπή. Πράγμα το οποίο πράξαμε, την αναθέσαμε εμείς. Έχουμε λοιπόν το τμήμα αυτό το υποκεφάλαιο Q στη διάθεσή μας. Βεβαίως, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, ένας χρόνος εμπειρίας δεν αρκεί για να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης, αλλά πάντως βλέπουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνέντευξη και συγκερασμό των πορισμάτων αυτού του υποτμήματος Q και των αποτελεσμάτων της έρευνας που έχει ανατεθεί. Έχουμε κανονιστικό έργο να ε, ξεκινήσουμε από εδώ και μπρος. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν αυτή τη στιγμή εκκρεμεί τη συζήτηση για το χρόνο πτήσεως, για τα όρια χρόνου πτήσεων, flight time limits, και σε διεθνές επίπεδο, όπως είπα και κατά την ομιλία μου, αλλά όπως θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από την κόπωση του πληρώματος κάτι το οποίο βαρύνει ιδιαίτερο ως προς τις ε, προδιαγραφές του χρόνου πτήσης, γιατί ο χρόνος πτήσης δεν είναι αυτός αυτός επικίνδυνος, όσο ο παράγων της κόπωσης των πληρωμάτων. Στους προσοχείς μήνες λοιπόν το θέμα αυτό θα το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Λαβάς νομίζω ήθελε κάποιο διαδικαστικό να υπογραμμίσει. Σύντομα, με ανησύχησε γιατί Όντω χρειάζεται να υπάρξει μια σαφή, ξεκάθαρη, διάφανη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων υπευθύνων. Έχω εδώ ένα κείμενο που μου έστειλε η Επιτροπή και όπου αναφέρει το ανάποδο από αυτό που είπε ο κ. Κουντού, ότι η Άσα έλαβε γρήγορα πρόσκληση από την Ισπανική Επιτροπή έρευνα του Τυχήματο, ότι έστειλε όλα τα στοιχεία που θεωρήθηκαν σημαντικά για την έρευνα, μεταξύ άλλων όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στον, ε, στο Μητρό Καταγραφή των Οργανωμένων Πτήσεως και ότι χορηγήθηκε το σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης της σχετικής έρευνας και ότι σχολιάστηκε πριν δημοσιευθεί. Η ισπανική δηλαδή προοπτική διαφέρει απόλυτα από τη δική σας δήλωση, σχόλιο τέλο πάντων, ότι η Επιτροπή, και αυτό είναι το μόνο με το οποίο συμφωνούμε κύριε Μπουντού, περιλαμβάνει ανεξάρτητους ερευνητές και από την κυβέρνηση και από τον κλάδο και από τον, ε, τις εταιρείες. Πάντω, αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι η Ισπανική Πεβέλα λέει ότι σα έδωσε ό,τι δυνατότητε ζητήσετε για να μπορεί να εμπλακείτε κι εσεί. ότι η πρόσκληση ξεκίνησε από την Ισπανία. Τέλο πάντων, ότι διευκολύναμε τη δουλειά. Σα ευχαριστώ και συγγνώμη. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε και μεταξύ μας λίγο. Όχι, όχι, λέει ο κύριος Γκουντού, δεν υπάρχει αντίρρηση. Λάβαμε τις πληροφορίες. Αυτό που είπα εγώ ήταν σχετικό με τα με το πρώτο τμήμα, τις πρώτες στιγμές, τις πρώτες μέρες της συνεργασίας. Εκεί καθυστερήσαμε. Στην αρχή ε, υπήρξε καθυστέρηση. Μετά βεβαίως ελήφθησαν όλα τα στοιχεία. Okay, well, again, thank you, Mr. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκουντού, λέει Πρόεδρος, για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας και ασφαλώς προσβλέπουμε σε πολύ καλή συνεργασία με τον οργανισμό σας. Όπως άλλωστε με όλους τους οργανισμούς με τους οποίους έχουμε συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα πάντως και για τους συναδέλφους ερωτώ. Εάν υπάρχει τίποτε άλλο στα διάφορα για την ημερήσια διάταξη, εάν όχι σημειώνω ότι στις 5 Οκτωβρίου στις 3.30 εδώ στις Βρυξέλλες θα διεξαχθεί η προσεχή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, και οι διερμηνείς ευχαριστούν και κυρίστε το πέρα στη